Καλημέρα, συνάδελφοι. Ξεκινάμε με την έγκριση της ημερήσιας ε, διάταξης. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνεται. Για τι γλώσσε θα έχουμε διερμηνία σε όλες, εκτός από την Κροατική, Δανέζικη και Ιρλανδική και περνάμε στις συστάσεις ε, των συντονιστών. Έχουμε ορισμό εισηγητών. Ρομπέρτα Μετσόλα έχει οριστεί εισηγήτρια για τον κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, η κυρία Σαρτζεντίνη των Πρασίνων για την οδηγία για τις κοινέ διαδικασίες ε, για την επιστροφή παρανόμως διαμενών των υπηκών τρίτων χωρών. Αυτά είναι τα μόνα. Εγκρίνονται, ωραία και μετά πάμε τώρα στις πράξεις ε, κάτω εξουσιοδότηση. Στις 3 Οκτωβρίου το Κοινοβούλιο έλαβε ένα σχέδιο απόφασης της Κομισιόν για το, το τμήμα του προγράμματος αξιολόγησης 2019 για την αξιολόγηση της Σέγγεν. Θα έχετε ενημερωθεί ήδη στις 5 Οκτωβρίου και η προθεσμία για αντιρρήσεις ε, ορίστηκε στις 17 Οκτωβρίου. Το βασικό νομοθέτημα είναι ο κανονισμός 1053 ε, του 2013 και βεβαίως έχουμε και ηλεκτρονική ψηφοφορία. Να έχετε λοιπόν παρακαλώ έτοιμες τις κάρτες σας. Οπότε έρχομαι στο πρώτο σημείο και χαίρομαι για το ότι έχουμε την παρουσίαση της έκθεσης για την αποστολή στην ΕΑΖΟ. Παρακολουθούσα εγώ στο Twitter, ήμουν σε άλλη αποστολή και ήταν πάρα πολύ σημαντική. Και είναι πολύ ενδιαφέρον οπωσδήποτε. Εισαγωγικά να σας πω Αυτό έχει μεγάλη σημασία και για τα προβλήματα εφαρμογής της νομοθεσίας στα κράτη πρώτης γραμμής και θα ακούσουμε από τον Πίτερ Νίντερ Μίλλερ και από άλλους ε, το τι κάνει η υπηρεσία. Έχουμε και τον ε, εκτελεστικό διευθυντή, τον προσωρινό, για να μας ενημερώσει για το τι κάνει η υπηρεσία. Νομίζω λοιπόν πρώτα απ' όλα θα ακούσουμε τον κύριο Αντού για να μας κάνει μια σύντομη παρουσίαση της υπηρεσίας ε, και κατόπιν ε, θα ακούσουμε και την αντιπροσωπεία. Η κυρία Άντερσεν ε, ήταν, είναι εδώ, όχι. Ποιο θα μας ενημερώσει τότε. Α, θα έρθει, μάλιστα. Η Μαρτίνα θα έρθει λοιπόν. Έχουμε τον κύριο Αντού. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, ξεκινήστε με την εισαγωγή σας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Χαίρομαι ιδιαίτερω ε, που είμαι εδώ πέρα μαζί σας σήμερα για να σας παρουσιάσω την ετήσια έκθεση του 2017 για την κατάσταση του ασύλου. Είναι ένα έγγραφο αναφοράς ε, που εκδίδεται ετησίως από το 2011 και χαίρομαι μπορώ να πω ότι έχετε εδώ πέρα τα πρώτα αντίγραφα. Τα λάβατε πριν από μένα μάλιστα. Και βεβαίως ε, έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο από το 2011. εστιάζει σε στατιστικά δεδομένα τη εξελίξη νομοθεσία, την πολιτική, την πρακτική και την νομολογία. Σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο μας λέει την πρακτική λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου και για εμάς είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στο να βρούμε κάποιους τομείς για βελτίωση και στήριξη και βεβαίως ε, μας δείχνει πού πρέπει να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας. Έχουμε λάβει λοιπόν συνεισφορές από τις εθνικές διοικήσεις, τα δικαστήρια, την κοινωνία των πολιτών, η πατερμοστία του ΟΗΕ, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και προσπαθήσαμε να κάνουμε μια ισορροπημένη ανάλυση της κατάστασης του 2017 και των ε, διδαγμάτων που έχουμε αντλήσει και μπορούμε να πούμε ότι φέτος λάβαμε συνεισφορές από 21 ε, οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών. Επόμενη διαφάνεια, ωραία. Πρώτα απ' όλα λοιπόν να σας δώσω κάποιες τάσεις του 2017 και για το 2018 και μετά θα πω τα κύρια σημεία. Πρώτα απ' όλα, έχουμε πάνω από 700.000 αιτήσει που υποβλήθηκαν το 2017, δηλαδή 44% λιγότερες από το 2016, μια σημαντική μείωση. Το 2017 είμαστε σε ένα επίπεδο ελαφρώς υψηλότερο από τα λεγόμενα επίπεδα προκρίσης του 2014, αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε στους πρώτους μήνες του 2018, επόμενη διαφάνεια, είναι ότι συνεχίζεται η τάση αυτή η πτωτική και έχουμε στο πρώτο εξάμεινο ένα 16% λιγότερες αιτήσει σε σχέση με το πρώτο εξάμεινο του 17. Ναι, ναι, αυτή ήταν η διαφορά σε σχέση με το 16. Βλέποντας τις χώρες προέλευσης, όπως για το 17 και το 18 Έχουμε Σύριους, Ιρακινούς και Αφγανούς, ε, τις κυριότερες εθνικότητες. Τούτων λεχθέντων βεβαίως πρέπει να σημειώσουμε ότι το 2017 οι Σύριοι υπέβαλαν πάνω από 108.000 αιτήσει ασύλου, ε, γύρω στο 70% λιγότερες από το 2016. Και αυτό ισχύει και αναλογικά για τους Ιρακινούς και Αφγανούς για να τα συγκρίνουμε. Έχουμε κάποιες ε, αυξήσεις από Βενεζουέλα, Γεωργία, Τουρκία και Κολομβία. Από αυτές τις χώρες αυξάνονται οι Τώρα, αν δούμε τις ε, λεπτομέρειες ανά κράτος μέλος, ελπίζω να φαίνεται η διαφάνεια, γιατί είναι μικρή η γραμματοσυρά. Περίπου τα μισά στα μισά κρατημέλη έχει μειωθεί ο αριθμό των αιτήσεων. Αρκετά σημαντικά. Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στην Γερμανία. Και ε, το βλέπετε αυτό. Έχουμε ε, πάει από τις 250 στις 800.000. Βλέπετε δεν είναι τελείως ε, στη σωστή κλίμακα και ο πίνακας. Έχουμε λοιπόν γύρω στις 500.000 λιγότερες αιτήσει που υποβλήθηκαν στη Γερμανία, οπότε η κατάσταση στη Γερμανία έχει ε, ένα σαφή αντίκτυπο στο σύνολο βεβαίως. Αν δούμε κάποιες συγκεκριμένες χώρες βλέπουμε ότι αντιθέτως στη Γαλλία οι αιτήσει αυξήθηκαν κατά το 1 πέμπτο, έφτασαν τις 100.000 και στην Ισπανία το 2017 διπλασιάστηκαν οι αιτήσει ασύλου κυρίως λόγω Βενεζολάνων που έρχονται χωρίς βίζα στην Ισπανία. Επόμενη διαφάνεια. Το 2018, το πρώτο εξάμεινο, η εικόνα είναι πολύ παρόμοια με λίγες εξαιρέσεις και ε, στη Γαλλία που ε, η αύξηση συνεχίζεται, η Ισπανία και η Κύπρος επίσης έχουν δει μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων σε σχέση με το 18 και έχουμε πολύ μεγάλη μείωση για την Ιταλία. Τις, με τις μισές ε, σχεδόν αιτήσεις. Επόμενη διαφάνεια. Να δούμε τώρα τις εκκρεμείς υποθέσεις. Ε. Εδώ πέρα εξετάζουμε τον αριθμό αιτήσεων που αναμένουν τελική απόφαση σε πρώτο επίπεδο ή σε δεύτερο. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων ε, είναι λιγότερος από το προηγούμενο έτος. Τούτου λεχθέντος έχουμε παρόλα αυτά σχεδόν ένα εκατομμύριο αιτήσει που εκκρεμούν στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου αν αναλύσουμε περαιτέρω τον αριθμό αυτό με τα δεδομένα της Eurostat και τα δικά μας. Να, αυτό είναι το 18, επόμενο. Βλέπουμε το τι γίνεται με τις αιτήσει σε πρώτο βαθμό. Αυτές μειώνονται αρκετά. Και επόμενο, αν συνυπολογίσουμε και όσες εκκρεμούν σε δεύτερο βαθμό, το κόκκινο κομμάτι, υπάρχει μια σαφής μετατόπιση της καθυστέρησης από τον πρώτο βαθμό στο δεύτερο βαθμό. Οπότε σε μεγάλο βαθμό έχουν κρυθεί σε πρώτο βαθμό οι αιτήσει του 2016 και οι αιτούντες αυτοί των οποίων οι αιτήσει απορρίφθηκαν εξακολουθούν να βρίσκονται μέσα στο σύστημα σε δεύτερο βαθμό και έτσι έχω την ευκαιρία να τονίσω ότι η ΕΑΖΟ στηρίζει και τα δικαστήρια από το 2013 και τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε εντείνει την στήριξή μας αριθμό εκπαιδεύσεων για δικαστές ε, και κάποια έγγραφα κατευθυντήρια για να υπάρξει μια σύγκληση των αποφάσεων σε δεύτερο βαθμό επόμενη διαφάνεια. Εδώ πέρα εξετάζουμε τον αριθμό των αποφάσεων που εκδόθηκαν και εδώ πέρα παρατηρούμε ε, γιατί έχουμε ακριβώ την μείωση των ακρεμών υποθέσεων παρά το ότι λοιπόν ο αριθμός ε, των ε, υποθέσεων αυτών είναι 40% αλλά ε, ο αριθμός των αποφάσεων είναι μόνο 13% μικρότερος. Βλέπουμε ότι οι προσπάθειες στα κράτη-μέλη ε, εντοπίστηκαν στην λήψη αποφάσεων 2017. Το 2017 οι μισές περίπου αποφάσεις ήταν θετικές. Αποφασίστηκε να δοθεί δηλαδή προστασία. Το 2018 που είναι το επόμενο slide παρατηρούμε ότι η τάση είναι παρόμοια με μία μικρή αύξηση των θετικών αποφάσεων που φτάνουν στο 40% περίπου των συνολικών ετοιμάτων για το πρώτο εξάμεινο του 2018. Η τελευταία γραφική παράσταση ε, είναι κατανομή αναχώρα προέλευσης. Αριστερά βλέπουμε τον αριθμό των που ελήθησαν για κάθε μία από τις χώρες και δεξιά ανατύπω απόφασης πρώτες τρεις χώρες αντικατοπτρίζουν με αντίστροφη σειρά και τον αριθμό των αιτημάτων. Θα δείτε τα δύο άκρα. Οι Σύριοι, για παράδειγμα, έχουν ένα μεγάλο αριθμό θετικών αποφάσεων, ευνοϊκών αποφάσεων, φτάνει στο 90%, ενώ οι Αλβάνοι είναι αυτοί που έχουν τους χαμηλότερους δείκτες αναγνώρισης. Στην ΕΑΣΟ ξεκινήσαμε πριν από τρία χρόνια μια διαδικασία για έκδοση κατευθύνων γραμμών αναχώρα. Ξεκινήσαμε το Αφγανιστάν συγκεκριμένα έτσι ώστε όλοι να έχουμε μια σχετικά κοινή εικόνα του τι σημαίνει στο Αφγανιστάν. Αυτό θα βοηθούσε τα κράτη-μέλη να τηρούν μια παρόμοια στάση σε σχέση με κάθε μία από αυτές τις χώρες. Περάμε στην επόμενη διαφάνεια. Ας δούμε ορισμένα συμπεράσματα από θεματικής πλευράς πλέον. Πρόσβαση στις διαδικασίες καταρχήν. Θα διαπιστώσουμε ότι η πρόσβαση στην επικράτεια των κρατών μέλων είναι μια βασική ανησυχία. Το αίτημα για διεθνή προστασία μπορεί να υποβληθεί σε αρχές του κράτους μέσα στην επικράτειά του ή στα σύνορα. Η κοινωνία των πολιτών αναφέρει ανησυχίες ό,τι αφορά τη δυνατότητα πρόσβασης λοιπόν στην επικράτεια με ένθερμο επιστροφές από πλευρά ενός αριθμού κρατών μελών, κάτι που αναφέρεται και από οργανώσεις δικαιωμάτων. Το 2017 άλλωστε αρκετές χώρες εξακολουθούν να ε, εφαρμόζουν την ε, προσωρι... τους προσωρινούς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Επίσης, η, διαδικα... η πρόσβαση στην διαδικασία ε, αποτελεί αντικείμενο ανησυχιών. Χρειάζονται νομικοί διάδρομοι για την πρόσβαση. Πάνω από 20.000 θεωρήσεις ε, ε, δόθηκαν για τη δημιουργία τέτοιων διαδρόμων από τη Γερμανία αλλά και από το Βέλγιο. Επίσης, ε, το 2016 εξαιτία τη σημαντική αύξηση των ετοιμάτων ε, πολλοί ετούντε ε, χρειάζονταν να περιμένουν ε, μεγάλο χρονικό διάστημα για να καταγραφούν. Αυτή τη στιγμή η το 2017 μια σημαντική βελτίωση της ταχύτητας. Αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι η υποδοχή και η καταγραφή να γίνονται στο ίδιο σημείο έτσι ώστε να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις. Για να μπορούν να επικοινωνούν πλήρως και για να καταλαβαίνουν και τα δικαιώματά τους οι ετούντες, χρειάζονται επαρκή και έγκαιρη πληροφόρηση. Όλο και περισσότερο οι κρατικές υπηρεσίες χρησιμοποιούν τι σύγχρονε τεχνολογίες και τα κοινωνικά δίκτυα για την παροχή πληροφοριών ή ακόμα και ε, εφαρμογές στα κινητά. Ένα άλλο θέμα είναι η διερμηνία, που είναι απολύτως απαραίτητη για την σωστή επικοινωνία των ετούντων με τις αρχές. Το 2017, κατά μέσο όρο, οι ευρωπαϊκές χώρες ε, έλαβαν αιτήματα από 54 χώρες σε σχέση με το 2016 είναι πολύ περισσότερο γιατί το 2016 ήταν μόνο 35 οι χώρες. Δηλαδή, οπότε σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες διερμηνίας οι προκλήσεις αυξάνονται. Χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερα τεχνολογικά μέσα όπως η τηλεφωνική διερμηνία ή η διερμηνία εξ ε, για την αντιμετώπιση των αναγκών νομική συνδρομή επίσης είναι σημαντική και το 2017 διαπιστώσαμε δύο ε, εξελίξεις προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Σε ορισμένα κράτη-μέλη ε, είδαμε την παγίωση και διεύρυνση ε, των, της νομικής συνδρομής όπως το Βελγίο ή τη Βουλγαρία. Κάποιες άλλες χώρες όμως έχουν ακριβώς την αντίθετη τάση όπως η Ουγγαρία για παράδειγμα τάση μείωση τη νομική συνδρομή που παρέχεται. Στην επόμενη διαφάνεια, εδώ θα δούμε ορισμένε σημαντικέ αλλαγέ στα εθνικά συστήματα. Πολύ δραστηριότητα σε νομοθετικό επίπεδο το 2017. Πολλά κράτη-μέλη δηλαδή τροποποιούν την νομοθεσία του. Αυστρία, Βέλγιο, Ουγγαρία και Ιταλία είναι μερικέ από αυτέ τι χώρε. Σε γενικές ε, γραμμές η προσπάθεια είναι να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος. Σε πολλά κράτη-μέλη δημιουργούνται διαδρομές για, για κάποιες κατηγορίες υποθέσεων. Αυτό σημαίνει ότι για καταφανώς αβάσιμες ή καταφανώς βάσιμες αιτήσει έχουν δημιουργηθεί πιο fast track διαδικασίες, πιο γρήγορες διαδικασίες για να ε, ολοκληρώνονται πολύ πιο γρήγορα. Οι ψηφιακές και άλλες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της ταυτοποίησης των ετούντων, οπότε βελτιώνεται και η ποιότητα της καταγραφής τους, πρώτη, τα πρώτα βήματα δηλαδή, της διαδικασίας. Πολλές χώρες επίσης έχουν ε, αυξήσει το, δυναμικό τους στη Φιλανδία, το Λουξεμβούργο, τη Σλοβακία και την Ελλάδα για παράδειγμα ε, με την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού. Ε, κατηγορία σε ασφαλών κρατών προέλευσης. Ε, έχει γίνει αναθεώρηση των, της ταξινόμησης. έξι κράτη-μέλη, για παράδειγμα, το 2017 εισήγαγαν τη Γεωργία ως ασφαλή χώρα προέλευσης. Επίσης παρατηρούμε αυξήσει επενδύσεων στους ε, μηχανισμούς αναθεώρησης των αναγκών προστασίας, έτσι ώστε να αφαιρείται η προστασία όταν πλέον δεν χρειάζεται συνθήκες υποδοχής. Συνολικά, το 2017 είδαμε μια μείωση της μεταναστευτικής πίεσης, της ε, πίεσης στην υποδοχή. Και κάποιες ε, πολλές χώρες μείωσαν τις ικανότητες υποδοχής τους, όπως για παράδειγμα το Βέλγιο, η Ελβετία, η Δανία, η Φιλανδία ή το Λουξεμβούργο, μειώνοντας τα κέντρα υποδοχής και τη χωρητικότητά τους. Επίση ε, πέρασαν σε πιο ε, σταθερές ε, εγκαταστάσεις, όχι προσωρινής φύσεως. Χώρες του Νότου όμως έχουν αυξήσει τις ικανότητές τους. Πορτογαλία, Ισπανία και Ιταλία είναι παραδείγματα τέτοιων χωρών. Να σας εντοπίσουμε ένα παράδοξο. Η ταχύτητα μείωσης των ικανότητων υποδοχής ακολουθεί τη μείωση των ετοιμάτων αλλά και τη μείωση των προϋπολογισμών. Αυτό ως παρενέργεια έχει την διατήρηση υψηλή πίεση στα κέντρα υποδοχή. δεδομένου βέβαια ότι έχουν μειωθεί τα κέντρα υποδοχή και η χωρητικότητά του. Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι σε ό,τι μας αφορά από το 2016 η υπηρεσία μας έχει επενδύσει σημαντικά σε έργο σχετικά με την υποδοχή, με ένα δίκτυο αρχών υποδοχής σε εθνικό επίπεδο. Όλες οι εθνικές αρχές αντιπροσωπεύονται εκεί. Αυτό οδηγεί σε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, καλύτερη συνεργασία. Αλλά επίσης έχουμε δημοσιεύσει και ένα αριθμό από έγγραφα, κατευθυντήρια έγγραφα, σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τις ε, προδιαγραφές που πρέπει να έχουν τα κέντρα υποδοχής και σκοπεύουμε να δημοσιεύσουμε και κατευθείαν μέσα για την υποδοχή παιδιών. Εξετάζουμε πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε την ποιότητα των προδιαγραφών των κέντρων υποδοχής σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Είναι σημαντικό επίσης να πούμε ότι η υποδοχή είναι ένα σημαντικό στοιχείο των δραστηριοτήτων στήριξής μας και σε όλα τα επιχειρημασιακά μας σχέδια στην Ιταλία, την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βουλγαρία μερικέ μερικές εβδομάδες έχουμε πολλές, πολλούς όρους, προδιαγραφές κλπ. για θέματα υποδοχής. Μέτρα για την βελτίωση της προστασίας των παιδιών. Η έγκαιρη, ο έγκαιρος εντοπισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ε, η ελλείψη έγκαιρου εντοπισμού ε, μπορεί να οδηγήσει στο να χαθούν τα παιδιά ε, και αυτό τα καθιστά θύματα, υποψήφια θύματα λαθρεμπόρων. Ένας αριθμός των μελών ανέπτυξαν ειδικέ υπηρεσίες υποδοχής παιδιών για να εξασφαλίσουν ένα περιβάλλον ασφαλές για τα παιδιά. Αλλά κράτη-μέλη βελτιώνουν ε, τη διαδικασία αξιολόγησης του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού ως τμήμα της διαδικασίας ασύλου. Εμείς υποστηρίζουμε τα κράτη-μέλη από την αρχή, από το 2011 που δημιουργηθήκαμε, υποστηρίζουμε τα κράτη-μέλη σε αυτό το θέμα. Να σας πω τι έχουμε κάνει, για παράδειγμα τι δημοσίευση έχουμε κάνει για αυτό το θέμα τελευταία. Έχουμε καταρχήν τον πρώτο οδηγό για την ε, εκτίμηση της ηλικία με διάφορες συστάσεις για το πώς πρέπει να γίνεται αυτή και σύντομα θα δημοσιεύσουμε, δημοσιεύσουμε ε, πρακτικές ε, συμβουλές για την, ε, ε, για την αξιολόγηση των παιδιών. Εστιάζουμε στα κράτη με πρώτης γραμμής, πέρσι για παράδειγμα, στηρίξαμε πολύ την Ιταλία σε σχέση με τους εφήβους. Εκεί στηρίξαμε την πρόσληψη και ε, επιμόρφωση εθελοντών φρουρών, ε, εθελοντών φροντιστών, συγγνώμη, που είναι πολύ σημαντικό. Αυτά. Τελευταία διαφάνεια ήταν αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Θα μπορούσα να συνεχίσω για πολύ χρόνο ακόμα, αλλά σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Θα ακούσω τις ερωτήσεις σας. Uh, ναι, ε, καθυστερήσαμε και να ξεκινήσουμε. Ε, δεν είχαμε αρκετά έγκαιρα αυτό το έγγραφο ε, για να σας το στείλουμε σε άλλους. Αλλά νομίζω πως όλα αυτά τα στοιχεία είναι πολύ χρήσιμα για τους συναδέλφους. Η Μαρτίνα λοιπόν ζήτησε το λόγο. Λέναντ, Νίντελ Μίλλερ... Λάμπερτ και η Μαρτίνα. Μαρτίνα πρώτα. Ναι, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Αλλά ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εισήγηση ε, και θέλω να ευχαριστήσω τον ε, Διευθυντή και το προσωπικό και να ευχαριστήσω και τη Γραμματεία αλλά και ε, την υπηρεσία της Μάλτας του Ευρωπαϊκού κοινοβούλιο για την διοργάνωση της επίσκεψής μας εκεί. Δεδομένου ότι η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από τη συνεχιζόμενη διαδικασία μεταμόρφωσης του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ασύλου σε ένα πραγματικό οργανισμό, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασύλου, είναι καλή ευκαιρία για να εξετάσουμε τον ισχύοντα και τον μελλοντικό ρόλο αυτού του οργανισμού. Αυτό οδήγησε σε μια μακροσκυλή συζήτηση για τη μεταρρύθμιση του οργανισμού αυτού μετά από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Ιουνίου που θα θυμάστε και μετά μέσα στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης μεταρρύθμισης του οργανισμού μετά από την ανανέωση του, ε, του προηγούμενου διευθυντή που, και του προσωπικού, του ανώτερου, του υψηλά ιστάμενου μάλλον προσωπικού, το οποίο συζητάσαμε με λεπτομερώς εδώ και ευχαριστούμε και τον Διευθυντή που μας αφιέρωσε αρκετό χρόνο. Η προσωπία μας ε, ε, μετέβη εκεί και συζήτησε πολλά θέματα όπως η στήριξη για το άσυλο, συμπεριλαμβανομένης ενημέρωσης, ανάλυσης, εκπαίδευσης, κατάρτισης των αρμοδίων στα κράτη-μέλη, δραστηριότητες σε τρίτες χώρες και το ε, πρόγραμμα ε, μετεγκατάστασης ε, ad hoc. Δεν μπορέσαμε να συζητήσουμε ειλικρινά και ανοιχτά μεταξύ μας και πραγματικά συγκεντρώσαμε πολλές, πολλές πληροφορίες και από την, νότα, τα τα στελέχη. Ε, μάθαμε από τις εμπειρίες ε, των προηγούμενων ετών. Εγώ θέλω να εκφράσω μια ανησυχία που δεν σχετίζεται με το την εργασία του ίδιου του, της ίδιας της υπηρεσίας ασύλου, αλλά αυτό που σας ζητά η Κομισιόν να κάνετε, που δεν ήταν σύμμορφο προς την ισχύουσα εντολή. Μάθαμε ότι πριν από περίπου έναν μήνα, ότι ζητήθηκε από το Γραφείο Στήριξης, από πλευράς της Κομισιόν, να δώσει πληροφορίες για πιθανές ασφαλείς τρίτες χώρες, δηλαδή ε, Βόρειος Αφρική, Δυτικά Βαλκάνια, Ουκρανία και Τουρκία. Είναι εξαιρετικά πολιτικού χαρακτήρα αυτό το θέμα και υπό την ισχύουσα νομοθεσία, τον ισχύοντα καθονισμό δεν ε, εμπίπτει στην εντολή, ε, την ισχύουσα εντολή του Γραφείου ε, Ασύλου. Θέλουμε εξηγήσεις από την Κομισιόν επ' αυτού. Μια παρατήρηση που νομίζω ξεπερνά αυτό το θέμα είναι ότι η Κομισιόν διαρκώς τροποποιεί το κείμενο. Μόλις ε, ολοκληρώσαμε όμως την διαπραγμάτευση. Δεν έχουμε, τώρα ξεκινάμε την εφαρμογή του και έχουμε την αίσθηση κάποιες φορές ότι είμαστε ε, σε, σε μέση εν, μιας μεγάλης, ενός μεγάλου εγχειρήματος δημοσίων σχέσεων που δεν βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες επιτόπου. Με τη νέα πρόταση για το Γραφείο Ασύλου ε, θα μπορέσουμε να προσφέρουμε επιχειρησιακή στήριξη σε όλες τις φάσεις ε, από τη συγκέντρωση στοιχείων ε, ιατρικών μέχρι τη φάση της έφεσης. Έχουμε και επιπλέον προϋπολογισμό ε, για προσωπικό, αλλά πιστεύουμε και φοβόμαστε πως αυτό θα οδηγήσει σε, μία απορρόφηση όλων αυτών των επιπλέον χρημάτων ε, ε, λόγω της τελέχωσης. Ενώ μια χώρα πρέπει να μπορεί να έχει τη στήριξη της υπηρεσίας αυτής όταν δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα ε, αιτήματα ασύλου όπως έχει γίνει στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Ε, Γι' αυτό και θέλω να συστήσω την προσοχή σε αυτό το θέμα. Βασικό δικαίωμα στο άσυλο θα πρέπει να προστατεύεται και να μην χρησιμοποιείται ως ένα εργαλείο για να επιταχύνονται οι επιστροφές. Το πολιτικό πλαίσιο εντό του οποίου γίνεται αυτή η πρόταση νομίζω μας δείχνει ότι ο στόχος αυτός μπορεί δυστυχώς να μην είναι ακριβώς ο στόχος της προστασίας αλλά να υπάρχει στόχος καταστολής και θα πρέπει βεβαίως να μελετήσουμε τις προτάσεις ε, μεταρρύθμισης ε, του, για, για τον οργανισμό αυτό και τις επιστροφές πράγμα που οδηγεί στην επιτάχυνση της διαδικασίας ασύλου και των επιστροφών στα σύνορα η Ευρωπαϊκή Επιρεσία Εξωτερικής Δράσης μέχρι που ζήτησε να υπάρξει παρακολούθηση για τις διαδικασίες διεθνούς προστασίας με πιθανές αποφάσεις επιστροφής σε περίπτωση αρνητικής ε, τελικής απόφασης. Πώς μπορεί αυτό να είναι σύμμορφο με την εντολή περί προστασίας και να πω ότι ορισμένοι εξημών στην αντιπροσωπεία βγήκαμε από την γραμμή και πήγαμε και επισκεφθήκαμε το Sea-Watch 3 και το πλήρωμά του. Επίσης ε, ε, επισκεφθήκαμε τα αεροσκάφη και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Μάλτα και όσοι έχουν διοριστεί εκεί ε, αντιμετωπίζουν. Ορισμένοι ήταν υπό νομική διαδικασία, άλλοι όχι και μπορέσαμε να, έτσι, να φωτίσουμε κάπως περισσότερο την κατάσταση εκεί και να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή στην επόμενη αντιπροσωπεία που θα επισκεφθεί τη Μάλτα. Και ξέρω πως αρκετοί συνάδελφοι εξέφρασαν ενδιαφέρον να αναγνωρίσουμε επίσης ότι ο Πίτερ Νίτερ Μιουλέρ που είναι σκιώδης της υπηρεσίας για το, σύνολο, για το άσυλο ήρθε μαζί μας και θέλω να εκφράσω την άποψή μου ότι θα έπρεπε να ήταν μέρος της επίσημης αντιπροσωπείας δεδομένου ότι είναι σκιώδης ε, δεν γίνεται να, να μην συμμετέχει δεδομένη της εμπειρίας του η συμμετοχή του και η παρουσία του εκεί εκτιμήθηκε από όλου όσοι, όσοι ήμασταν εκεί. Θέλω να ευχαριστήσω τη Γραμματεία και είμαι βέβαιος, βέβαια μάλλον, ότι και οι υπόλοιποι που δεν είχαν την ευκαιρία να έρθουν θα μελετήσουν την έκθεσή μας ε, από αυτή την αποστολή. Ευχαριστώ πολύ Μαρτίνα για την ε, εμπεριστατωμένη σου αυτή αναφορά. Ορισμένοι μιλήσατε για την πρόταση της Κομισιόν προς την Επιτροπή, ε, προς την, ε, μάλλον τον οργανισμό, ε, που είναι το επόμενο θέμα. Και φυσικά θα το συζητήσουμε πλήρως. θέλω να ελέγξω τώρα αν υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που συμμετείχαν σε αυτή την αντιπροσωπεία. Ο Πίτερ, μετά η Άννα και μετά η Μπιργκίτ. Και ο Τεϊρόν επίσης που ήταν μέλος της αντιπροσωπείας. Πίτερ. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Αντού και την, το επιτελείο του γιατί όλοι γνωρίζουμε πως το γραφείο αντιμετώπισε κρίση και κατάφερε να διαχειριστεί με εξαιρετικό τρόπο την κρίση αυτή και μπορούμε αυτό να το δούμε και με βάση αυτή την παρουσίαση ότι δηλαδή η ΆΖΟ εργάζεται πολύ αποτελεσματικά μετά από την κρίση που ε, διένυσε και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας. Ήθελα να το πω εξ αρχή Δεύτερον, η Μαρτίνα ήδη ανέφερε και νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ακόμα μια φορά πως η ΕΑΖΟ χρειάζεται οπωσδήποτε περισσότερο προσωπικό. Όχι μόνο χρήματα και κόσμο, ανθρώπους. Γιατί λεφτά χωρίς ε, ανθρώπους δεν έχει νόημα. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να, να γίνουν τα απαραίτητα βήματα σε αυτό το τομέα. Ε, Επίση είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ε, τη σημασία της κατάρτισης. Γιατί με την επίσκεψή μας στη Μάλτα πραγματικά πήραμε μια πολύ εντυπωσιακή παρουσίαση για τη ε, διαδικασία της δραστηριότητα μάλλον εκπαίδευσης ε, εκεί στην ΕΑΖΟ και είναι πάρα πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη να το κάνουν αυτό. Τελευταία μου παρατήρηση για την παρουσίαση, κυρία Αντού. Νομίζω πως είναι σαφές πως έχουμε όλο ένα και λιγότερη ε, ε, προσήλωση. Και ξέρω πως τα κράτη-μέλη μιλάνε για τη μεταναστευτική πίεση και τι θα κάνουμε κτλ. Και, και το άσυλο. Έχουμε λιγότερες αιτήσει αλλά περισσότερη πολιτική ιστορία. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι το σύνολο της μεταναστευτικής πολιτικής της Ένωσης και της προσφυγικής πολιτικής της Ευρώπης έχουν πέσει, γίνει όμοιροι πολιτικών χειρισμών και αυτό δεν έχει να κάνει με τη δραστηριότητα της ίδιας της ΕΑΖΟ. Θα πρέπει να εξετάσουμε το πολιτικό πλαίσιο εντός το οποίο γίνεται αυτή ε, η συζήτηση. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ξεκάθαρα στατιστικά στοιχεία για να ξέρουμε ακριβώς ποια είναι η κατάσταση και ότι δεν μπορεί να συγκριθεί με την κατάσταση του 2015 ή του 2016. Σας ευχαριστώ πολύ. Επειδή ήθελε και ο κύριος Λέναρτς, αλλά πείτε μας εσείς πρώτα, γιατί ήσασταν και εσείς στην αντιπροσωπεία. Πάντα, πάντα σύντομα κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει ο κύριος Λέναρτς για την επίσκεψη της αντιπροσωπείας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και ευχαριστώ τον κύριο Αντού και όλο το προσωπικό για την φιλοξενία και το εξαιρετικό πρόγραμμα. Όπως είπε και ο Πίτερ ε, όλοι γνωρίζαμε για την κρίση. Δεν, ξέρω το, δεν ξέραμε τι έπρεπε να περιμένουμε πηγαίνοντα εκεί, αλλά εγώ θεωρώ ότι βρήκαμε μια υπηρεσία που στεκόταν στα πόδια της. Έχουμε πραγματικά ανθρώπους, επαγγελματίες, που προσπαθούν να αποκαταστήσουν πρώτα απ' όλα την φήμη της υπηρεσίας ε, και ζητούσαν βεβαίως περισσότερους πόρους, περισσότερο προσωπικό γιατί αντιλαμβάνονται ότι η φήμη και η αξιοπιστία της υπηρεσίας πρέπει να αποκατασταθεί και χρειάζονται πόροι γι' αυτό και πρέπει εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και συμφωνώ με αυτό το οποίο είπε και ο Πίτερ. Το θέμα δεν είναι μόνο λεφτά, αλλά ανθρώπινοι πόροι και προσωπικό στην ε, ΕΑΖΟ, ειδικά δει κανεί τι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Μιλώντας για τις προκλήσεις αυτές, ε, έχουμε εγώ έχω διαφορετική αίσθηση για την πίεση που υπάρχει, γιατί πράγματι υπάρχουν λιγότερε αφήξει. Ε, τώρα δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι έχει τελειώσει η κρίση. Είχα μια συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα που πολλοί ομιλητέ λένε ότι ε, το θέμα είναι πια πολιτικό, γιατί τα στατιστικά αισθία λένε ότι δεν υπάρχουν πια ε, τόσο πολλέ αφήξει. Αλλά το σημαντικό είναι ο αριθμό των εκκρεμών υποθέσεων και το τονίσατε αυτό, βλέπετε, για το 2017. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει η κατάσταση. Ε, υπάρχει ουσιαστικά ένα εκατομμύριο ε, υποθέσεις που εκκρεμούν ακόμα. Εντάξει, ίσως να είναι διαφορετικό είδος ε, κρίσης, πρόκλησης, όπως θέλει να το πει κανείς, αλλά η πίεση στο σύστημα ασύλου των κρατών μελών ε, είναι βεβαίως κάτι το οποίο αξίζει προσοχής ε, και νομίζω ε, ήταν σαφές αυτό και στην σημερινή παρουσίαση γιατί βεβαίως είναι κάπως περίεργο να μιλάμε για το 2017, ειδικά αν έχετε και τα στοιχεία του 2018, ίσως και του Σεπτεμβρίου ακόμα. Σας ευχαριστώ λοιπόν και αναμένω την περαιτέρω συνεργασία στο μέλλον. Ευχαριστώ Μπιργκίτ. Θα εστιάσω σε μία ερώτηση εγώ ε, σε σχέση με αυτό το οποίο είπε ο κύριο Λένα για το 1 εκατομμύριο εκκρεμεί υποθέσεις και να λέμε ότι αυτό είναι άλλου είδου πίεση προ τα κράτη-μέλη. Αναρωτιέμαι γιατί 1 εκατομμύριο έχουμε 520 εκατομμύρια πολίτες έχουμε ένα εκατομμύριο εκρεμής υποθέσεις ε, είναι η πίεση και σε ποιες χώρες. Νομίζω ότι τις περισσότερες από αυτές ε, ε, είναι σε δύο-τρεις χώρες, οπότε τα περισσότερα κράτη-μέλη δεν έχουν αυτή την πίεση. Και πρέπει να το τονίσουμε και αυτό. Από την άλλη, ίσως οι χώρες όπου δεν έχουν αυτή την πίεση έχουν τη μεγαλύτερη καταστολή και δεν θέλουν να εργαστούν πάνω σε αυτό το θέμα. Και έτσι έρχομαι στη δεύτερη μου ερώτηση, γιατί κύριε Διευθυντά αναφέρατε τις συνθήκες υποδοχής ε, που σε κάποιες χώρες ε, ε, χειροτερεύουν. Ποιες είναι αυτές οι χώρες και πόσους ετούντες έχουν πέρσι ή φέτος και μπορείτε να μας πείτε με ποιον τρόπο ακριβώς αυξάνεται η πίεση όσον αφορά τις συνθήκες υποδοχής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Άννα. Ευχαριστώ κύριε Αντού για την πολύ σημαντική παρουσίασή σας ε, και τα σημαντικά στοιχεία που πραγματικά δεν ταιριάζουν με την ρητορία που συνεχίζει συνεχίζουν κάποιοι που έχουν κακούς σκοπούς. Αναφέρατε τις ανησυχίες ε, της κοινωνίας των πολιτών που μιλάνε για ανθρωπιστικούς διαδρόμους ε, και ανθρωπιστικές αποστολές. Νομίζω ότι εμείς συμφωνούμε με αυτά. Αλλά οι ε, ανθρωπιστικοί διάδρομοι είχαν νόημα όταν είχαμε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης όπως στην Συρία το 2015 και πιο πριν Και βεβαίω περιγράψατε ότι οι Σύριοι, οι Ιρακινοί, οι Αφγανοί είναι οι περισσότεροι ετούντε. Ε, δεν θα είχε νόημα η ΕΑΖΟ να ανοίξει εγκαταστάσει σε χώρε όπω η Ορδανία, η Αίγυπτος, ο Λίβανος, η Τουρκία για να γίνει εκεί μια επεξεργασία των αιτήσεων. Για να μην περιμένουμε δηλαδή να ε, έρθουν παρανόμως χωρίς έγγραφα, χωρίς βίζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να υποβάλουν αίτηση. Και τέλος, ε, δεν ξέρω αν ε, τα κράτη-μέλη συνεχίζουν να είναι επιλεκτικά όσον αφορά τη μετακατάσταση, γιατί ξέρουμε ότι συνέβη αυτό στο παρελθόν. Ο κόσμος ήθελε μόνο χριστιανούς, ε, ξανθούς κτλ. σε κάποια κράτη-μέλη. Και ε, ζητώ συγγνώμη, δεν θα ακούσω την απάντησή σας. Αλλά κάποιος θα τα ακούσει. Γιατί πρέπει να πάω κάπου αλλού, κάτι το οποίο δείχνει την υποκρισία των κρατών μελών. Ε, γιατί ασχολούνται με τους μετανάστες αλλά ανοίγουν ε, γρήγορα τις αγκαλιές τους πλούσιους μετανάστες γιατί μπορούν να πληρώσουν χρυσές βίζες και δίνουν ε, μέσως ε, υπηκότητες ε, και έτσι διαστρεβλώνεται η Σέγγεν. Σας ευχαριστώ. Θα συζητήσουμε τις προτάσεις κομισιών αργότερα, οπότε θα φτάσουμε σε αυτό. Θα ήθελα να ζητήσω από τον κ. Αντού να απαντήσει ιδιαίτερα στις αρχικές παρατηρήσεις κ. Σάντερσον, αλλά και στα υπόλοιπα. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Καταρχήν, να ευχαριστήσω και την αντιπροσωπεία που μας επισκέφθηκε. Δεν δεχόμαστε συνήθως τόσο μακρές επισκέψεις, διήμερες. Συζητήσαμε σε βάθος πάρα πολλά πράγματα και με Πάντοτε με χαρά δεχόμαστε επισκέπτες, αλλά συνήθως δεν μένουν για παραπάνω από δύο ώρες. Προσπαθούμε να τους ενημερώσουμε σε ένα πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αυτή τη φορά η επίσκεψη ήταν ε, διήμερη, χρήσιμη πολύ για μας, ελπίζω και για σας. Δεν θα σχολιάσω τις νέες προτάσεις της Κομισιόν, μια και είναι το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Αλλά να πω για τα υπόλοιπα. Ασφαλείς χώρες. Σίγουρα δεν είναι τμήμα της εντολής μας να αξιολογήσουμε το κατά πόσον μια τρίτη χώρα είναι χώρα ασφαλής. Αλλά να σας ξεκαθαρίσω ότι οτιδήποτε κάνουμε εμπίπτει στην εντολή μας. Δηλαδή δίνουμε πληροφορίες για τις χώρες προέλευσης. Δεν κάνουμε καμία αξιολόγηση. Είναι αντικειμενικές, αμερόληπτες και ουδέτερες πληροφορίες για τις τρίτες χώρες. Άλλοι θα τις αξιολογήσουν και θα βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Ευχαριστώ πολύ τα μέλη της αντιπροσωπείας για τη στήριξή τους, τη στήριξη του έργου μας. Προσπαθούμε ασφαλώς να ανακτήσουμε την αξιοπιστία της, ε, του οργανισμού μας, της υπηρεσίας μας. Σε ό,τι ε, το καλοκαίρι ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα δράσης για τη διακυβέρνηση αξίας με 53 μέτρα. Δεν θα σας αναφέρω λεπτομέρειες. Το συζήτησα και με την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού του Κοινοβουλίου τον περασμένο μήνα. Το, ο στόχος όλων αυτών είναι η αξιοπιστία, να βελτιωθεί η αξιοπιστία. Και εδώ Σίγουρα θα συνεργαστούμε με όλους τους εταίρους μας, μεταξύ αυτών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενισχύουμε τους εσωτερικούς μας ελέγχους και, την... και τις μας. Με αύξηση του προσωπικού είναι μεγάλη ανησυχία για μας. Θέλουμε να αυξήσουμε το προσωπικό μας κατά 30% μέχρι την αρχή του χρόνου όπως ακριβώς είχε προβλεφθεί από το οργανόγραμμά μας. Επίσης, γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να δώσουμε χέγγια για να γίνουμε πιστευτοί και αξιόπιστοι. Η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου αναφέρει ότι χρειάζομαστε περισσότερο προσωπικό όχι μόνο για να επιτελέσουμε το έργο μας, αλλά και για να ε, μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τις υποχρεώσεις μας σε σχέση με, το, με την ε, εκτέλεση του προπολογισμού μας. Ε, εξελισσόμαστε από κέντρο ειδικευμένη γνώσης σε κέντρο ειδικευμένη γνώσης και στήριξης πρώτης γραμμή, οπότε χρειαζόμαστε να έχουμε ειδικευμένο προσωπικό και για αυτό τα, τα καινούργια καθήκοντά μας. Βέβαια, οτιδήποτε γίνει θα πρέπει να σέβεται τους δημοσιονομικού κανόνες και τους κανόνες διαφάνειας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την υποδοχή. Δεν μιλούσα για τις συνθήκες υποδοχής, αλλά για τις ικανότητες και το, τη χωρητικότητα των κέντρων υποδοχής. Αυτό που είπα είναι ότι αυτές οι ικανότητες μειώθηκαν, αλλά η πίεση εξακολουθεί να παραμένει. Λετωνία, Λιθουανία, Ισπανία και Πορτογαλία έχουν ανοίξει καινούρια κέντρα υποδοχής, οπότε έχουν αυξήσει την, τις ικανότητές τους, αλλά άλλες χώρες τις, έχουν μειώσει. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, έχει αυξηθεί ο αριθμός των αιτήσεων πάρα πολύ, ενώ στην Ιταλία έχει μειωθεί σημαντικά. Οπότε είναι δύσκολο να βγάλουμε συμπεράσματα για τις συνθήκες και για την πίεση που δέχεται κάθε χώρα. Ε, το θέμα της ε, κατάρτισης και της επιμόρφωσης ε, δεν αποτελεί αντικείμενο αυτής της έκθεσης, αλλά η εκπαίδευση, η επιμόρφωση ήταν πάντοτε τμήμα του έργου μας. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Σχολείο Ασύλου για τους ε, υπαλλήλους ε, πρώτου βαθμού αλλά και για δικαστές. Πάνω από 26.000 άτομα έχουν ήδη συμμετάσχει από το 2012 στα σεμινάρια επιμόρφωσης που οργανώνουμε. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το έργο αυτό. Είναι πολύ σημαντικό και για να εξασφαλίσουμε μια ενιαία αντιμετώπιση των ετούντων. Θέλουμε ένα κοινό παρανομαστή με τις ίδιες πληροφορίες, με τις ίδιες διαδικασίες, με την ίδια γλώσσα σε εισαγωγικά. Θέλουμε όμοιες πρακτικές. Τέλος, για τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους και την εμπλοκή της ΑΣΟ ε, στο μέλλον. Αυτά έχουν, οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι έχουν ε, μια εξωτερική διάσταση με πολύ σημαντικά νομικά προβλήματα, αλλά αυτό δεν θα τα σχολιάσω. Απλά να πω ότι η, η ΑΣΟ παίζει, έχει να παίξει σημαντικό ρόλο στην επανεγκατάσταση. Πριν από δύο εβδομάδες μάλιστα ξεκινήσαμε ένα σχέδιο στην Τουρκία για ένα μηχανισμό στήριξης της επανεγκατάστασης για τα κράτη-μέλη. Ε, και ελπίζουμε στις αρχές του 2019 να έχουμε μια πιλωτική εκατάρτιση για να δούμε πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τη δράση μας αυτό το θέμα στο μέλλον. Νομίζω ότι κάλυψα τις περισσότερες ερωτήσεις. thank you very much, uh, Mr. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αντού. Και όπως είπαμε έχουμε την πρόταση της ε, Κομισιόν που θα συζητηθεί μετά. Οπότε θα δούμε κάποια από αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστήσω την αντιπροσωπή για την επίσκεψη τέσσερις αντιπροσωπείες νομίζω της ΛΥΜΕ ε, ταξίδευαν εκείνη την εβδομάδα. Δηλαδή ε, θα πρέπει ακριβώ να δούμε αυτό το, το θέμα. Να δούμε το τι γίνεται στα λόγω κράτη και οι αρμόδιοι πάλι να είναι έμπειροι και βεβαίως ε, και οι βουλευτές μας εδώ πέρα αποκτούν εμπειρίες και αυτό επηρεάζει νομοθεσία. Ήταν λοιπόν αρκετά καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε. Σας ευχαριστώ κυρία Ντού. Ξέρω πως θα συναντηθείτε και με άλλους συναδέλφους είναι μια στιγμή ευαίσθητη για την υπηρεσία σας. Περνάμε τώρα στην παρουσίαση της ε, Κομισιόν ε, για τον κανονισμό του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο. Λοιπόν, ε, είχαμε επιτύχει μια πρώτη συμφωνία τον Ιούνιο του 2017 επί Μαλτέζικης Προεδρίας, οπότε τώρα η συμφωνία πρέπει να ξανανοίξει και δεδομένου του ότι η πρόταση αυτή βεβαίως δεν είναι μόνη της αλλά σχετίζεται με την προσωρινή συμφωνία του Ιουνίου 2017 η Επιτροπή μας αποφάσισε να δημοσιεύσει αυτή την προσωρινή συμφωνία και μπορείτε να την βρείτε στα έγγραφα της σημερινής συνεδρίασης με την συμφωνία βεβαίως και των άλλων δύο θεσμικών οργάνων. Δεδομένης λοιπόν της ε, σημασίας της μεταρρύθμισης του συστήματος ε, ασύλου η Επιτροπή μας αποφάσισε να δει αυτήν την πρόταση με βάση το επιτυχημένο χρονοδιάγραμμα και μόνο στα αγγλικά. Οπότε αναφέραμε πριν το ότι ο εισηγητής της ΛΥΜΠΕ είναι εισηγητής ε, για αυτήν την πρόταση, είναι ο κύριος Νίτερ Μίλλερ θα δώσω λοιπόν τον λόγο στον Πίτερ για να μας πει κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα όμως ε, θα ζητήσουμε την Κομισιόν να κάνει μια παρουσίαση της πρότασης αυτής. Και θα ζητήσουμε από τον κύριο Ράιαν να μας κάνει μια πρόταση, ο οποίος είναι τμήματάρχης αρμόδιος για το θέμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. στις 12 ε, Σεπτεμβρίου η Κομισιόν ενέκρινε ένα πακέτο μέτρων, τρεις στοχευμένες προτάσεις και μια ανακοίνωση με στόχο να ενισχυθεί η ικανότητα της Ένωσης να διαχειριστεί τη μεταναστευσή όπως εξήγησε και ο πρόεδρος Γιούνκερ την ίδια ημέρα. Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος ε, όσον αφορά τη δημιουργία ενός πιο του πλαισίου, αλλά απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες έτσι ώστε η Ένωση να έχει τις δυνατότητες να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει συγκεκριμένα. Θα πρέπει να επιτευχθούν συμφωνίες ε, για ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου που θα βρίσκει την σωστή ισορροπία μεταξύ αλληλεγγύης και ευθύνης και μια ισχυρή ευρωπαϊκή τέτοια υπηρεσία είναι βασικός πυλώνας ε, του Ευρωπαϊκού Κοινού Συστήματος Ασύλου και ένα βασικό μέσο αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν τέτοιες πιέσεις. Μία ενισχυμένη τέτοια υπηρεσία θα πρέπει ακριβώς να παρέχει όλη την τεχνική αρρωγή που χρειάζονται τα κράτη-μέλη, να συνεργάζεται ακόμη στενότερα με τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες για να υπάρχει μια ολοκληρωμένη απάντηση. Γι' αυτό η Κομισιόν έχει υποβάλει στοχευμένες αυτές ε, αλλαγές στην αρχική της πρόταση. Σκοπεύουμε να υπάρχει μια σαφώς καθορισμένη νομική εντολή για όλες τις επιχειρησιακές ε, δραστηριότητες που πιθανώς ε, θα κληθεί να υλοποιήσει και δεν θα πρέπει βεβαίω να μπορεί να στηρίξει τα κράτη-μέλη με οποιονδήποτε τρόπο απαιτηθεί. Θα ήθελα να τονίσω πω η τροποποιημένη αυτή πρόταση σέβεται πλήρω την προσωρινή πολιτική συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των συνομοθετών πέρσι τον Ιούνιο του 2017 συγκεκριμένα. Επί της αρχής πρότασης της Κομισιόν του Ιουλίου η νέα πρόταση βασίζεται σε αυτή την προσωρινή συμφωνία και λαμβάνει υπόψη τις ε, εμπειρίες των τελευταίων δύο ετών, ειδικά στην Ελλάδα και την Ιταλία. Μάλιστα αυτές οι εμπειρίες έδειξαν ότι πρέπει να επεκτείνουμε ακόμη περισσότερο την επιχειρησιακή και τεχνική αρρωγή που παρέχει η υπηρεσία στα κράτη-μέλη. Οι στοχευμένες τροπολογίες που περιέχονται εδώ, σε συνδυασμό με τις ε, προτάσεις που υιοθετήθηκαν την ίδια ημέρα για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Νοριακής και Ακτοφυλακής και ευθυγράμμιση της οδηγίες περί επιστροφών. Όλες αυτές οι αλλαγές νομίζω και θα πρέπει να τονίσω είναι περιορισμένες και θα πρέπει να θεωρούνται συμπληρωματικές προς τα όσα έχουν ήδη συμφωνηθεί. Λοιπόν, για να δούμε συγκεκριμένα τις λεπτομέρειες των όσων έχουμε προτείνει. Στόχος είναι τα κράτη-μέλη να έχουν ενισχυμένη στήριξη από την υπηρεσία για να μπορούν να επεξεργάζονται τις αιτήσει για διεθνή προστασία γρήγορα και γέρος μέσω της διευκόλυνσης της εμπλοκής της υπηρεσίας σε όλες τις πτυχές της διαδικασίας στο διοικητικό στάδιο και στην ε, διαδικασία κρίσης του ποιο κράτος μέλος είναι υπεύθυνο σύμφωνα με τον κανονισμό Δουβλίνου και στην ε, δυνατότητα διοικητικής αρρωγής στην φάση των ε, δευτεροβάθμιων προσφυγών και βεβαίως μπορεί να δοθεί στήριξη στα κράτη-μέλη μόνο κατόπιν ετοιματός τους, δεν θα επιβάλλεται σε αυτά. Επιπλέον, πρέπει να τονίσουμε πως η τελική απόφαση είτε σε πρώτο βαθμό είτε σε δεύτερο βαθμό πάντα είναι αρμοδιότητα των εθνικών αρχών και η ακριβής σύνθεση του πακέτου στήριξης πάντα θα προσαρμόζεται στις ανάγκες των κρατών μελών σε ένα επιχειρησιακό σχέδιο. Η πρόταση επίσης έχει στόχο να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ της Υπηρεσίας Ασύλου και της υπηρεσία συνοριοφυλακή ε, Θα συνεργάζονται ήδη αυτές οι υπηρεσίες ε, και από κοινού θα μπορούν ε, να αναπτύσσουν ομάδες στήριξης αντιμετώπισης της μετανάστευσης για να αντιμετωπίσουν όλες τις προκλήσεις που έχουν τα κράτη-μέλη. Τρίτον, η πρόταση προβλέπει την ανάπτυξη αυτών των ομάδων όχι μόνο σε καταστάσεις δυσανάλογης πίεσης, όπως είχαμε πέρσι το καλοκαίρι, αλλά και ως ένα προληπτικό εργαλείο με στόχο καλύτερης διαχείρισης των μεικτών μεταναστευτικών ροών που ζουν τα κράτη-μέλη. Και σύμφωνα και με την τρέχουσα πρακτική σε Ιταλία και Ελλάδα προβλέπουμε επίσης ότι ο γενικός συντονισμός των ομάδων αυτών πρέπει να ανοίξει στην Κομισιόν και αυτό τώρα έχει διευκρινιστεί στις προτινόμενες ε, τροπολογίες και αλλαγές της εντολής. Αυτό διασφαλίζει συνοχή, οικονομία πόρων και συνέργεια μεταξύ των διαφόρων δράσεων. Όλες αυτές οι αλλαγές βεβαίως συμμορφώνονται με την ε, πρόταση που καταθέσαμε την ίδια μέρα ε, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και άρα θα ενισχυθούν δύο υπηρεσίες. Τέταρτον, προτείνεται να ευθυγραμμιστεί το πλαίσιο διοίκησης με την κοινή προσέγγιση για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Ιουλίου 2012, ένα πλαίσιο το οποίο είχε συμφωνηθεί μεταξύ Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Κομισιών, όπως γνωρίζετε και αυτό το οποίο έχουμε συγκεκριμένα αλλάξει, προτείνει να αλλάξει είναι να δοθεί στην Κομισιόν η ευθύνη να προτείνει υποψηφίους για τον αναπληρωτή εκτελεστικό διευθυντή για να ισχύει η ίδια διαδικασία που προτείνουμε και για τον εκτελεστικό διευθυντή. Επίσης, μια ανάλογη αλλαγή προτείνεται και στην Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή. Και τέλος, για να ολοκληρωθεί η αποστολή με αυτήν την ε, διευρυμένη έντολη, προτείνονται και 55 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον κονδύλια μεταξύ του 2019 και 2027. Έτσι θα υπάρχει δυνατότητα να αναπτύσσονται σχετικές ομάδες όπου απαιτείται με τον κατάλληλο αριθμό ειδικών, τεχνικού εξοπλισμού και υποδομών και μια που έχουν ήδη γίνει κάποιες ερωτήσεις, ε, ήδη από τον κύριο Νίντερ Μίλλερ και την κυρία Άντερσον ε, μπορώ να εξηγήσω το γιατί δεν προτείναμε ταυτόχρονα επιπλέον ανθρώπινους πόλους. Να πω πρώτα απ' όλα ότι απαιτούνται ανθρώπινοι πόροι για την υπηρεσία Βεβαίω είχε σοβαρή αύξηση του προσωπικού τα τελευταία χρόνια, κάτι το οποίο συνεχίζεται, αλλά δεν νομίζαμε ότι ήταν ε, απολύτως αναγκαίο να προβλέψουμε επιπλέον προσωπικό για να μπορεί η υπηρεσία να κάνει την δουλειά της με βάση τη διευρυμένη εντολή. Και υπ' αυτήν την έννοια πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι τα επιπρόσθετα κονδύλια σε έναν σημαντικό βαθμό θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση ειδικών στην σύνθεση των ομάδων που θα αναπτύσσονται. Και τέλος, καλώς ορίζουμε το γεγονός ότι η Επιτροπή αποφάσισε να χρησιμοποιήσει ένα επιταχυμένο χρονοδιάγραμμα για την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Ράιν, πολλά μας είπατε και για τον εισηγητή και για τους άλλους ε, συναδέλφους. Και... Ως γενικό σχόλιο θα ήθελα να πω ότι όλοι θέλουν να δουν ποια θα είναι η πραγματική πραγματικά, πραγματική προσθέμενη αξία γιατί όλοι ανησυχούν για την αξιοπιστία της υπηρεσίας. Θα δώσω τώρα στον κύριο Νίντερ Μίλλερ, που είναι ο εισηγητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που αυτό το θέμα το θέσατε, στην, το βάλετε στην ημερησία διατάξη. Είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να ευχαριστήσω και την Κομισιόν για την παρουσίαση και για την προετοιμασία αυτού του θέματος, αυτού του φακέλου. Τον Μάιο του 2016, όπως όλοι γνωρίζουμε, η Κομισιόν μαζί με άλλες προτάσεις υπέβαλε και μια πρόταση κανονισμού για την, τον, Ευρωπαϊκ, τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άσυλο. Ο στόχος ήταν ε, η, ο οργανισμός αυτός να αποκτήσει τις, ε, τα μέσα που χρειάζεται για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ε, των, μεταναστών και των προσφύγων. Ή ο οργανισμός θα έπρεπε να λειτουργήσει το συντομότερο δυνατό. Οι διαπραγματεύσει δεν ήταν απλές, αλλά καταφέραμε να καταλήξουμε σε πολιτική συμφωνία με το Συμβούλιο το καλοκαίρι του 2017. Το κείμενο αυτής της πολιτικής συμφωνίας ε, δημοσιεύθηκε στο, στη σελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, και είναι διαθέσιμο. Η πολιτική αυτή συμφωνία για μας εξακολουθεί να ισχύει και με εκπλήσει που το Συμβούλιο δεν είναι ικανό να βρει μια, ένα συμβασμό για αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα. Οπότε οι προτάσεις Κομισιόν με εκπλήσουν γιατί όχι μόνο ανοίγουν την αρχική προσωρινή συμφωνία των συνομοθετών αλλά αλλάζουν και το ίδιο το περιεχόμενο με καινούρια καθήκοντα που παρέχονται στον οργανισμό. Ε, ενώ το Δουβλίνο ακόμα τελεί υπό διαπραγμάτευση. Τι γίνεται με το, με το νομικό στάτους της προηγούμενης συμφωνίας. Από ό,τι ακούω η, συμφων... η, η Κομισιόν συμφωνεί με την προσωρινή συμφωνία του 2017, αλλά αν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε η κατάσταση είναι πραγματικά θολή. Δεν καταλαβαίνω τις προθέσεις αυτής της καινούρια πρότασης, αυτών των καινούργιων προτάσεων. Σύμφωνα με τη δική μας αξιολόγηση, όλες οι προτάσεις της Κομισιόν που έχουν ως στόχο την βελτίωση της σύνδρομης θα μπορούσαν να γίνουν στο πλαίσιο και κάτω από την ομπρέλα της προσωρινής συμφωνίας. Οπότε χρειάζεται να τις διαπραγματευτούμε. Όπως αναφέραμε στην Αυστριακή Προεδρία, μεταξύ μας υπάρχει πλήρη συμφωνία ε, μεταξύ δηλαδή και των εισηγητών και των συσκιωδών εισηγητών όλων των πολιτικών ομάδων απόλυτη συμφωνία να μην γίνει καμία επαναδιαπραγμάτευση ε, των προσωρινών συμφωνιών των προηγούμενων ετών. Αυτό ήταν πολύ σαφής και ξεκάθαρη δήλωση των εισηγητών και συνεισηγητών. Η πρόταση της Κομισιόν μάλιστα μας δημιουργεί και διαδικαστικά ζητήματα που δεν τα έλαβε υπόψη η Κομισιόν όπως γνωρίζω. Συμβουλευθήκατε το Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία και το πώς θα διαρθρωθεί αυτή πριν υποβάλλετε τις προτάσεις σας. Προφανώς μας ενδιαφέρει η αύξηση του προπολογισμού του οργανισμού, απολύτως απαραίτητη, αλλά μία ακόμα φορά να πω ότι λυπούμαστε που δεν, προβλέπονται, που δεν προβλέπεται αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού. Η αύξηση του προπολογισμού χωρίς αύξηση του προσωπικού δεν έχει πολύ νόημα. Ε, συνοψίζοντας, πρέπει να πω ότι δεν νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να τροποποιήσουμε την πολιτική συμφωνία στην οποία είχαμε καταλήξει το καλοκαίρι του 2017 σε συνεργασία με το Συμβούλιο. Αυτή είναι μια γενική άποψη ε, όλων των εισηγητών και των σκιωδών εισηγητών. Ευχαριστώ. Θα μας... Θα θα συζητήσουμε τα θέματα, τα διαδικαστικά, τα νομικά και του προσωπικού, αλλά ας ακούσουμε πρώτα τους Κιώδης εισηγητής. Ο κ. Κοέλιο, από το ΕΛΚ. Συμφωνώ με τον κύριο Νίτερ Μίλλερ. Υπενθύμησε ότι το καλοκαίρι του 2017 υπό Προεδρία της Μάλτας, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε μια προσωρινή συμφωνία για τη νέα νομική βάση του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο. Από τότε, μια σειρά άλλων προσωρινών συμφωνιών επετεύθηκαν για μηχανισμούς σχετικούς με το άσυλο. Όλα αυτά μπλοκαρίστηκαν στο Συμβούλιο. Τώρα φαίνεται ότι η Κομισιόν θέλει μαζί με το Συμβούλιο να καθυστερήσει ακόμα περισσότερο ε, την υιοθέτηση των προσωρινών συμφωνιών. Α το δούμε προσεκτικά. Η Κομισιόν υποβάλλει μια πρόταση που απαιτεί μια άλλη πρόταση η οποία ήδη έχει αποτελέσει αντικείμενο προσωρινής συμφωνίας. Αλλά ας δούμε και την ουσία της πρότασης που υποβάλλει η Κομισιόν. Επιτρέπει να συγκλίνουν οι δύο συνομοθέτες, δημιουργεί μια πιο ευέλικτη νομική βάση για τον νέο οργανισμό, έτσι ώστε να υλοποιήσει καλύτερα το τροποποιημένο ε, σύστημα ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυξάνει τις αρμοδιότητες και τις ικανότητες του μελλοντικού οργανισμού. Δυστυχώς η απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα είναι ένα εκοφαντικό όχι. Εξ όσων γνωρίζω, Έχουμε μια συμφωνία στο τραπέζι. Διαθέτουμε συμφωνία. Και από όσο γνωρίζω, ήταν αυτό ήταν το πρώτο θέμα το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο προσωρινή συμφωνία πάνω από ένα χρόνο πριν. Δεν γνωρίζουμε ποιε είναι οι προθέσεις τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αυτή την πρόταση. Δεν γνωρίζουμε τι θέλει το Συμβούλιο. Αλλά γνωρίζω, είμαι σίγουρο για το τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να εγκρίνουμε το νέο οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άσυλο και πριν το τέλος της θητείας μας μάλιστα. Θέλουμε να πετύχουμε αυτό το στόχο. Ο εισηγητής, ο Πίτερ Νίντερμιλερ, μπορεί να είναι σίγουρος για την στήριξή μας έτσι ώστε να εγκριθεί η υπάρχουσα συμφωνία χωρίς καθυστέρηση. Ενίσχυση λοιπόν της θέσης ε, του εισηγητή ήσασταν σαφής και κάθετος. Το ακούει και η Πρόεδρια. Είμαι βέβαιος ότι παρόμοια θα είναι και η θέση των υπολείπων σκιωδών. Μαρτίνα. Ναι, εγώ θέλω να συμφωνήσω με το όσο είπε ο Πίτερ και πρέπει να πω πως κάπως έχω μείνει άναυδη. Γιατί η Κομισιόν φαντάζομαι πως καταλαβαίνει τα ωφέλη του να έχουμε, μία, να έχουμε ένα μακροχρόνιο εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο εργάζεται για ένα συγκεκριμένο θέμα, ειδικά όταν πρόκειται για τέτοιο θέμα. Και ε, πρέπει λαπή, κατά συνέπεια να, να, καταλάβει και να συμπεράνει ότι θα περιλαμβεί εκεί επιπλέον ε, καθήκοντα και αύξηση του προϋποσωπικού, αλλά ε, θεώρησε ότι δεν μπορούσε να ε, αυξήσει το προσωπικό γιατί μπορεί να προσλαμβάνει ειδικούς εξωτερικούς συνεργάτες. Όταν όμω θέλει κανεί να φτιάξει πυρογνωμοσύνη, όπω φαντάζομαι πώ το κάνει και η Κομισιόν μέσα στην ίδια τη λειτουργία τη, τότε θα έπρεπε να καταλαβαίνει καλύτερα τι χρειάζεται ένα τέτοιο οργανισμό. Και απορρίπτω παντελώ αυτή την έννοια ότι δηλαδή μπορεί να αναθέτει όλο ένα και περισσότερα καθήκοντα, να αυξήνει τον προπολογισμό, αλλά να λε ότι δεν πειράζει. Θα προσλαμβάνω για μικρά διαστήματα πυρογνώμονε, ανθρώπου που πάνε και έρχονται εντάξει, με καλές προθέσεις και με ειδικέ γνώσεις, αλλά που δεν μπαίνουν μέσα σε αυτήν την ε, δομή ώστε να μπορέσουν να ε, ε, εμπεδώσουν εκεί και να παγιώσουν την εμπειρογνωμοσύνη τους. Απλώς μετακινούνται μαζί με την εμπειρογνωμοσύνη τους από δεξιά και αριστερά. Επίσης θέλω να ρωτήσω αν η Κομισιόν μπορεί μαζί μας να μοιραστεί τη διατύπωση του αιτήματο που προήλθε από την Κομισιόν που ε, ενήργησε μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ασύλου για πιθανές τρίτες χώρες, ασφαλείς τρίτες χώρες. Εμένα με εξεκολουθεί να με προβληματίζει αυτό παρά τα όσα είπατε και ίσως κάτι που θα μπορούσε να ελαφρύνει την ανησυχία μου εάν δεν υπάρχει βάσιμη αν θεωρείτε μάλλον πως δεν είναι βάσιμη η ανησυχία μου. Θέλω να ακούσω λοιπόν όχι απλά εκφράσεις και λόγια, αλλά να μας δώσετε ένα αντίγραφο του τι στείλατε στο Ευρωπαϊκό ε, Γραφείο Στήριξης για το Άσυλο. Πράγμα το οποίο, όπως είπα, θα άρει τις ανησυχίες μου αυτές. Ευχαριστώ. Οι υπόλοιποι σκιώδεις δεν μπορούσαν να είναι παρόντες, αλλά νομίζω πως ε, εν γέννη καταλάβαμε το νόημα. Ε, υποστηρίζεται η θέση του εισηγητή. Θα στραφώ και πάλι λοιπόν στην Επιτροπή και θα ζητήσω από τον Σάιμον Πράμερ της Αφυσιακής Προεδρίας να πάρει το λόγο. Επίσης έχουμε δύο μήνες ακόμα και θα ήθελα κάπως έτσι ευθαρσώς να ρωτήσω αν μπορείτε να μας πείτε τι συμβαίνει με αυτή τη δέσμη για το άσυλο γενικότερα. Τι άλλες πληροφορίες μπορείτε να μας δώσετε, αν μπορείτε γιατί και αυτό θα μας βοηθήσει για τα συγκεκριμένα νομοθετικά ζητήματα που έθεξε ο εισηγητής. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Νίντερ Μίλλερ, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην Επιτροπή σας ε, και για την δυνατότητα που μας δίνετε να μιλήσουμε. Ευχαριστώ και την ε, Κομισιόν για την υποβολή της ε, τροποποιημένης ε, πρότασης, η οποία όπως ακούσαμε ήρθε στις 12 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστώ και τον Στίβεν. Ε, επιτρέψατε μου πρώτα απ' όλα να αντιδράσω σε κάποια από αυτά τα οποία ακούστηκαν, έχοντας βεβαίως κατά νου ότι και για εμάς και την Προεδρία είναι σαφές ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίζεται στην προσωρινή ένωση, στην προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθη με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί Μαλτέζικης Προεδρίας, οπότε δεν σκοπεύουμε να αποκλίνουμε από το συμφωνημένο κείμενο. να σας πω τώρα το πώς ακριβώς ε, είδαμε αυτή την ανακοίνωση Κομισιόν στις 12 Σεπτεμβρίου να σας ενημερώσω ότι είχαμε μια πρώτη εξέταση αυτής της πρώτης της Κομισιόν ήδη στις 25 Σεπτεμβρίου ήδη αυτή την ε, εβδομάδα στις 8 Οκτωβρίου είχαμε μία νέα συνεδρίαση στο επίπεδο του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών όπου είχαμε τις πρώτες συμβιβαστικές προτάσεις που τις οποίες υποβάλαμε και η επόμενη διαβούλευση όπως είπα θα γίνει πάλι στο επίπεδο του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών στις 26 Οκτωβρίου. Σκοπεύουμε λοιπόν να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις, ε, να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν ε, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει η αναλογή πλειοψηφία. Χαίρομαι που ακούω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σκοπεύει να προωθήσει το θέμα στην Επιτροπή σας ε, με την ε, επιταχυμένη διαδικασία και ευχαριστώ τον κύριο Νίντερ Μιούλερ, τον εισηγητή, για την συνεργασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Um, ευχαριστώ. Τι να κάνουμε τώρα. Mr. Ryan, do you want to add to our um, Κύριε Ράιν, εσείς έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο έτσι, στην γενική μας κατάθλιψη. Ε, τέλος πάντων, συγγνώμη, έχετε να πείτε τίποτα. Να επανέλθω στο θέμα. Ακτός αν θέλει ο το γιατί νομίζω ότι όλοι είμαστε έτσι κάπως. Κάπως πεσμένοι. Λοιπόν, ε, για το θέμα των επιπλέον πόρων ε, το απάντησα. Εμείς δεν θεωρούσαμε ότι ήταν ε, αναγκαίο ειδικά δεδομένου του ότι στην τρέχουσα πρόταση προτείνεται να αυξηθεί το προσωπικό στα 500 άτομα, μια πολύ σημαντική αύξηση σε σχέση με σήμερα και δεν θεωρούσαμε ότι απαιτείται κάτι περαιτέρω. Αλλά σημειώθηκαν αυτά τα οποία είπαν οι βουλευτές ε, σήμερα. Όταν μιλάμε για την προστιθέμενη αξία, αυτά τα οποία είπαν ο κύριος Νίντερ Μιλέρ και ο κύριος ε, Κοέλιο, αυτό το οποίο μπορώ να κάνω εγώ είναι να επαναλάβω ότι πρόκειται για πολύ στοχευμένες ε, τροπολογίες και αλλαγές. Δεν έχουν στόχο να ανοίξουν τις ευαίσθητες ε, πτυχές του κειμένου που είχε συμφωνηθεί το καλοκαίρι θεωρούμε ότι αυτές οι αλλαγές ε, μπορούν να γίνουν χωρίς να ξανανοίξει κάτι από αυτά τα ευαίσθητα ε, θέματα και συγκεκριμένα θα επισήμενα το ότι η αρχική πρόταση της Κομισιόν έγινε το καλοκαίρι του 2016. Είχαμε σημαντική πειρά τα δύο χρόνια που πέρασαν εν τω μεταξύ ειδικά με την στήριξη που παρέχει η υπηρεσία στα hot spots σε Ελλάδα και Ιταλία και βεβαίως αντλήσαμε εκεί τα διδάγματά μας και είπαμε ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει περαιτέρω η εντολή. Ταυτόχρονα θεωρήσαμε ότι είναι αναγκαίο να διασφαλίσουμε ότι οι ομάδες αυτές στήριξης θα μπορούσαν να πτήσονται σε διάφορες περιπτώσεις σε πολύ περισσότερες σε σχέση με την προσωρινή πρόταση και άρα πρέπει να δούμε τις αλλαγές που προτείνονται στην συνοριοφυλακή και ότι για να λειτουργήσει σωστά θα έπρεπε να γίνονται κάποιες αλλαγές στην εντολή της υπηρεσίας ασύλου και κάτι τελευταίο ο προϋπολογισμός όπου όπως τονίσατε ο επιπρόσθετος προϋπολογισμός απαιτείται και αυτή είναι νομίζω μια αλλαγή που κάνει η τροποποιημένη πρόταση. Αυτό που είπε η κυρία Άντρισον για πληροφορίες για ασφαλείς τρίτες χώρες το καλύψατε. Θέλετε να πείτε κάτι. Uh, για τις ασφαλείς τρίτες χώρες. Πράγματι μας ζητήθηκε, ζητήθηκε από την ΕΑΖΟ να κάνει κάποια έρευνα για πιθανές υποψήφιες χώρες για έναν κατάλογο ασφαλών τρίτων χωρών Αυτό είναι κάτι το οποίο είχε ζητήσει το Συμβούλιο. Και αντιλαμβάνομαι ότι είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ κύριε Ράιν. Ναι, χαίρομαι που απαντήσετε. Θα, θα έβγαζα ένα συμπέρασμα ακόμη πιο καταθλιπτικό, αλλά πείτε αν έχεις εσύ κάτι να πεις, ίσως να είναι καλύτερο από αυτό που θα πω εγώ να απαντήσω και εγώ στο τέλος αν υπάρχουν άλλα σχόλια. Αν θέλει κάποιος άλλο βουλευτής να πει κάτι. Μαρτίνα, ένα, ένα πράγμα. Ε, ξέρω πως αυτό το οποίο λέει η Κομισιόν ε, ισχύει. Θέλω ακριβώ οι βουλευτές να έχουν τη φύση του αιτήματο. Δηλαδή να μας στείλετε το τι ζητήθηκε και πώς ζητήθηκε πράγματι το έχετε επιβεβαιώσει, το γνώριζα ούτως ή άλλως. Δεν είναι... Δεν είναι θέμα επιβεβαίωση. Θα ήθελα να δω ακριβώς το τι ζητήθηκε από την ΕΑΖΟ. Την αλληλογραφία, email ότι ήταν... Αν μπορείτε να το στείλετε στους βουλευτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ θα επανέλθω. να είναι ναι, σαφές αυτό. Και Πίτερ, θέλεις να πεις κάτι σύντομα να πω και πάλι ένα ευχαριστώ στην Κομισιόν για την απάντηση και την πρόταση. Και τώρα θα μιλήσω γερμανικά και βεβαίως χαίρομαι ε, όταν ακούω πως η Αυστριακή Προεδρία θέλει να κάνει τις διαπραγματεύσεις γρήγορα. Εγώ είμαι πάντα στην διάθεσή σας και θα χαιρόμουν να κινηθούμε το συντομότερο δυνατόν γιατί θεωρώ ότι όλοι εντός της αιθούσης συμφωνούν στο ότι θεωρούμε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Σύλλου ένα πολύ σημαντικό μέσο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Και ακριβώ χρειαζόμαστε αυτή τη στήριξη από την Αυστριακή Προεδρία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ράιεν, για το συγκεκριμένο θέμα αυτό που έθιξε η κυρία Άντερσον, θέλετε να απαντήσετε. Ναι, σύντομα. Προφανώς δεν έχω το κείμενο μπροστά μου προτείνω να έρθουμε σε επαφή με την γραμματεία κάποια στιγμή να δούμε ε, αν μπορούμε να σας δώσουμε περαιτέρω λεπτομέρειες. Ναι, ναι, καλώς, θα το, θα το δούμε. Ναι, κατανοητό αυτό το οποίο είπε ο εισηγητής. και πραγματικά θέλετε να συναντηθούν οι συντονιστέ για να δούμε τα όσα λέει η Κομισιόν γιατί δεν είναι ικανοποιητικά και υπάρχει μια πολιτική συνένεση από αυτού. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το δούμε στο πλαίσιο του πακέτου. Γι' αυτό ζήτησα από την... Ρώτησα την Προεδρία αν μπορεί να μιλήσει για αυτό το θέμα. Βλέπω εδώ πέρα ότι πραγματικά αγανακτούν, αλλά και εμείς αγανακτούμε, γιατί όλα αυτά είναι συνδεδεμένα και εσείς έχετε τον δικό σας ε, κύβο του Ρούμπικ, το αντιλαμβάνομαι. Πρέπει να το δείτε σε αυτό το πλαίσιο στην ε, συνάντηση των συντονιστών. Γιατί θα πρέπει να υπάρξει κάποια αλλαγή στο πακέτο, κάποια κίνηση στους τελευταίους δύο μήνες. Ας δούμε λοιπόν το τι θα γίνει. Αλλά από την δική μας την ε, πλευρά υπάρχει πολιτική συνένεση για την ε, νομοθετική προσέγγιση. Ευχαριστώ λοιπόν τους εισηγητές, οι σκιώδες θα συναντηθούν οπωσδήποτε και θα μας πούν. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ και την Προεδρία συνάδελφοι, περνάμε τώρα στο σημείο 6, πρόγραμμα δικαιώματα και αξίες. Εδώ πέρα θα ακούσουμε την παρουσίαση του προγράμματος για την περίοδο 2021 2027. Όπως ξέρετε, η πρόταση αυτή αφορά τους στόχους και τον <coughs> προπολογισμό του προγράμματος και βεβαίω αφορά τους κανόνες της με το νέο πρόγραμμα περί δικαιοσύνης θα αποτελέσει τμήμα του προϋπολογισμού της ΕΟΚ για να έχουμε ανοιχτές, πλουραλιστικές και δημοκρατικές κοινωνίες. Τον λόγο έχει λοιπόν ο εισηγητής. Παρακαλώ, αν δεν θέλετε να αποχωρήσετε λίγο ήσυχα Κυρία Μπόντι. Σε τα και πρώτα Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω ειδικά, μια και μου δίνεται αυτή η ευκαιρία. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους και εισηγητές και τους άλλους ε, εισηγητές. Το θέμα αφορά πολλές διαφορετικές επιτροπές. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, και όλες τις οργανώσεις ε, με τις οποίες ήρθα σε επαφή ε, τα τελευταίο καιρό, την Επιτροπή των Περιφερειών. Το θέμα είναι τι συμβαίνει τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορισμένες από τις αρχές πάνω στις οποίες έχουμε βασίσει όλο το οικοδόμημα αυτή τη στιγμή αμφισβητούνται ή και καταπατούνται, αγνοούνται σε ορισμένα κράτη-μέλη. Και μάλιστα, από ό,τι φαίνεται, οι πολίτες δεν είναι και πολύ καλά ενημερωμένοι για το ποια είναι τα δικαιώματά τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον Απρίλιο του 2018 υιοθετήσαμε ένα ψήφισμα για αύξηση του ποσού των οργανώσεων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων και οργανώσεων κοινωνία των πολιτών που εργάζονται σε, σε θέματα δικαιωμάτων, αρχών και αξιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή στηρίζουμε οργανώσεις, πολλές οργανώσεις και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που δραστηριοποιούνται στο θέμα των δικαιωμάτων αλλά δεν στηρίζουμε με τον ίδιο τρόπο οργανώσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό αποφασίσαμε τον, τον Απρίλιο και η Κομισιόν υπέβαλε μια πρόταση και χαίρομαι που το έκανε. Με την πρότασή της διευρύνει το πεδίο υφιστάμενων προγραμμάτων έτσι ώστε αυτά να μπορέσουν να καλύψουν περισσότερα θέματα που έχουν σχέση με το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, χωρίς όμως να αυξήσει τα ποσά το οποίο σημαίνει ότι προγράμματα τα οποία ήδη υπάρχουν και υποχρηματοδοτούνται θα πρέπει να καλύψουν ένα πιο ευρύ φάσμα θεμάτων. Ήδη ακόμα και έτσι όπως είναι η κατάσταση, η κοινωνία των πολιτών λέει ότι δεν χρηματοδοτούνται παρκώς αυτά τα προγράμματα. Τώρα πώς είναι δυνατόν με τα ίδια χρήματα να χρηματοδοτήσουμε και περισσότερες δράσεις. με τους σκιώδεις εισηγητέ προσπαθούμε να καθορίσουμε την θέση του Κοινοβουλίου. Οι περισσότεροι από τους σκιώδεις συμφωνούν με τις προτάσεις οποίες υποβάλλει. Οι προτάσεις μας έχουν να κάνουν καταρχήν με το πεδίο εφαρμογής. της πρότασης. Δεν θέλουμε οι καινούριε προτάσεις να βλάψουν τα υφιστάμενα προγράμματα. Γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε ένα καινούριο πυλώνα που θα βασίζεται στο άρθρο 2 και τις, ε, που θα αφορά μάλλον το άρθρο 2 και τις θεμελιώδεις αρχές της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης προτείνουμε μια αύξηση του προπολογισμού έτσι ώστε να καταστεί αυτό δυνατό. Αν δεν αυξηθεί ο προπολογισμό, τότε τα καινούρια, τα ήδη φυστάμενα προγράμματα θα δουν να του τραβάνε το χαλί κάτω από τα πόδια. Επίσης, θέλουμε να αυξήσουμε την συμμετοχή των πολιτών στην δημοκρατική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 500 εκατομμύρια ευρώ είναι ένα ευρώ αναπολίτη. Αυτό που ζητάμε είναι το 40% των ποσών αυτών να φτάσει εγγυημένα όμως στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Ορισμένες περιφέρειες και τοπικές αρχές ήδη το κάνουν, συγγνώμη, ήδη ασχολούνται με θέματα δικαιωμάτων, κράτους δικαίου κλπ. Αλλά είναι πολύ σημαντικό οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να έχουν δυνατότητα να απορροφήσουν αυτά τα κονδύλια. Αυτή τη στιγμή οι οργανώσεις οι οποίες δεν είναι διεθνείς ε, και είναι απλώς ε, εσωτερικού βελνικούς μέσα στο κράτος μέλος δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση από αυτά τα προγράμματα. Χρειάζεται επίσης να χρηματοδοτούνται και ε, και η οργάνωση κοινωνία των πολιτών, δηλαδή έχουν μια βασική χρηματοδότηση που να μην σχετίζεται με συγκεκριμένα προγράμματα. Πρέπει λοιπόν να διευκολύνουμε το ρόλο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Και η Κομισιόν το προσπαθεί στην ε, πρότασή της. Ένα από τα ζητήματα που προκύπτουν είναι το ότι κάθε σημείο επαφής θα πρέπει, που πρέπει να υπάρχει στα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο ε, η ψηφοφορία θα λάβει χώρα στις 10 Δεκεμβρίου. Και οι τροπολογίες μπορούν να κατατεθούν μέχρι τις 26 Νοεμβρίου. Είμαι σίγουρη ότι θα συνεργαστούν πολύ καλά. Ευχαριστώ. Um, Σε ευχαριστώ πολύ, Μποντίλα, για αυτή σου την εισήγηση. Σκιώδης τώρα για το ΕΛΚΑ. First of all, Ο κύριος ε, ε, Μπόνι, με συγχωρείτε. Ε, καταρχάς να σας ευχαριστήσω για το σχέδιο και τη δική σας προσπάθεια γιατί είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω πως από κοινού μπορούμε να καταστήσουμε αυτό το, το φάκελο ρεαλιστικό στην εφαρμογή. Ευχαριστώ που λάβατε ένα, που περιλάβατε μάλλον ένα κομμάτι του ψηφίσματος στην πρόταση τώρα. Ε, πιστεύω και αισθάνομαι κάποιο αν, μάλλον ε, δεν αισθάνομαι απόλυτα ικανοποιημένο, γιατί έχουμε στηρίξει βέβαια τις ανάγκες ε, των οργανισμών σε τοπικό επίπεδο βέβαια, αλλά πιστεύω πως πρέπει να αλλάξουμε το πεδίο εφαρμογή και να εστιάσουμε περισσότερο στις ε, τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, να είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο, στην ε, άσκηση της δημοκρατίας, ε, της διδαχής, της συμμετοχικής Τη συμμετοχής μάλλον στη δημοκρατία, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το μέλλον της. Έπειτα θα πρέπει να υπάρξει και αποσαφένιση κάποιων κανόνων. Βεβαίω, όλα θα πρέπει να είναι διαφανή, ε, αλλά να δούμε και ποιο είδος μοντέλο θέλουμε, όπως ανέφερε η Μποντίλ Βαλέρο, η διεθνής διάσταση θα το καταστήσει αυτό πολύ πιο θετικό και χρήσιμο για τις ε, ε, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι όταν μιλάμε για το πρόγραμμα αξιών έχουμε δεξιότητες και δικαιώματα, οι πολίτες και συμμετοχή και αυτός και το πρόγραμμα Δάφνη που είναι πολύ σημαντικό στην πρόληψη της βίας κατά των παιδιών, των νέων και των γυναικών. Και συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση τη συζητήτρια ότι δηλαδή χρειάζεται να έχουμε μια ειδική ε, πτυχή ε, ξεχωριστά για την Ένωση, γιατί θα είναι έτσι πιο εύκολο να οργανώσουμε τις δραστηριότητες με διαφανή τρόπο ε, προς τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Τελευταία παρατήρηση σχετίζεται με τον προϋπολογισμό. Περιμέναμε 1,5 δις για αυτό το μέσο, όπως λεγόταν πριν. Τώρα, όταν κανείς αναλύσει τα προγράμματα σε αυτό το τίτλο «Επένδυση στον κόσμο», βλέπουμε πως το, Ευρωπαϊκό, Κοινωνικό Ταμείο παραμένει στην ίδια, στο ίδιο επίπεδο. Το Erasmus Plus αυξάνεται, το European Solidarity Corps ε, επίση 200% αύξηση. Η Δημιουργική Ευρώπη αύξηση. Άλλα προγράμματα αύξηση. Οι αποκεντρωμένες ε, νεοργανισμοί αύξησης. Αλλά όταν δούμε δικαιώματα, δικαιοσύνη και αξίες, μείον 8 είμαστε σε σύγκριση με τα προηγούμενα προγράμματα. Πράγμα που δείχνει πως έχουμε πρόβλημα με τους πόρους. Συμφωνώ με την πρόταση της εισηγήτριας ότι θα έπρεπε να είναι το κονδύλι πολύ υψηλότερο σε σύγκριση με την πρόταση που παρουσίασε η Κομισιόν, όμως από την άλλη πλευρά Έχω κάποιες αφιβολίες για το αν θα είναι δυνατό να συζητήσουμε με τους συναδέλφους ε, τον προϋπολογισμό. Πιθανώς λοιπόν να πρέπει να σκεφτούμε εάν το προτινόμενο επίπεδο 1,5 δις με, τις, με το κομμάτι το χωριστό για τις αξίες θα πρέπει να αυξηθεί βέβαια σε συνεργασία με τις άλλες επιτροπές και την Επιτροπή Προπολογισμού, αλλά έχουμε κάποιο χρόνο για τροπολογίες. Και τέλος να προσθέσω κάτι ακόμα, διότι νομίζω πως χρειάζεται να κατανοήσουμε πόσο σημαντικά είναι αυτά όλα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για όλους μας. Το να στηρίξουμε δηλαδή τις ε, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ειδικά σε σχέση με τις εκθέσεις που συντάσσει η Επιτροπή Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που δείχνουν όσο πολύ συρρυκνώνεται η δραστηριότητα των ε, οργανώσεων των πολιτών. Δεν είναι θέμα πολιτικής ιδεολογίας, είναι ουσιώδες για να ενταθεί η συμμετοχή όλων των πολιτών από όλες τις χώρες ώστε να έχουμε μια ισχυρή δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Σκιώδη για το Σοσιαλιστέ είναι η Σεσίλ Κέγκε. Παρακαλώ, Σεσίλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Κλοντ. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την ε, μεγάλη δουλειά ε, τροποποίησης που έχει ήδη κάνει. Είχαμε ήδη την ευκαιρία να συναντηθούμε, να συζητήσουμε και εξ ονόματο τη ομάδα των σοσιαλιστών μπορώ να πω πω οι τροπολογίε σα ε, βρίσκουν σύμφωνους ε, απόλυτα και προχωρούν προς την κατεύθυνση που είχαμε αρχικά υποδείξει στην αρχή αυτή της διαδικασία, γιατί στηρίζονται και προωθούνται οι ευρωπαϊκέ αξίε, αλλά και η έννοια της ηθαγένεια. Θα πρέπει πιστεύω να σταθούμε σε αυτό, να αυξήσουμε και να προωθήσουμε την έννοια της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Με χαρά λοιπόν δέχομαι την αλλαγή του τίτλου του προγράμματος, όπου περιλαμβάνεται και η Ιθαγένεια, καθώς και την επέκταση του πεδίου εφαρμογή του κανονισμού και στο τμήμα αξίες της Ένωσης, όπου δεν μπορούμε φυσικά να ξεχνάμε το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία που είναι σημαντικά στοιχεία απαραίτητα για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ένωση. Συμμερίζομαι με την εισηγήτρια την ανάγκη διεύρυνση των μορφών προστασία στα τμήματα που ήδη υπάρχουν και αναφέρομαι συγκεκριμένα τη στήριξη που δίνεται στα θύματα της βίας για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, καθώ και άλλε προσθήκες στην καταπολέμηση των διακρίσεων και των αντι ε, να ενημερώσω δε την συγκήτρια ότι θα υποβάλω τροπολογία για την αφρικανοφοβία μια φοβία απέναντι στους ανθρώπους που προέρχονται από την Αφρική και η οποία αντίνεται όλο και περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, θα μιλήσω για τον ε, γραφειοκρατικό φόρτο, γιατί πρέπει να εγγυηθούμε τη δυνατότητα πρόσβασης στα προγράμματα τα ευρωπαϊκά και των μικρών οργανώσεων. Επίσης, ε, θα πρέπει να ενθαρρύνουμε διάλογο των ε, ε, των ε, οργανώσεων των πολιτών με ε, την ευρωπαϊκή δομή. Θα πρέπει επίσης να μιλήσουμε για δομές στήριξης για τους δικαιούχους των προγραμμάτων. Ωστόσο, να είμαστε κάπως περισσότερο ευέλικτοι. Σε πολλές χώρες μέλη αυτές οι δομές υπάρχουν ήδη. Οπότε, θέλουμε να τις ενισχύσουμε ή να τις χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να μην υπάρξουν επικαλύψεις. Τέλος, η χρηματοδότηση. Όπως ήδη είπε ο συνάδελφος Μπόνιλ, η συνάδελφος Μπόνιλ, υπάρχει σημαντική αύξηση του κονδυλίου, αλλά όχι επαρκής για το δικό μας τομέα, γιατί οι προκλήσεις είναι πολυάριθμες για τις ε, οργανώσεις των πολιτών που καταπολεμούν την ξενοφοβία, την παρότρινση σε μίσος. Ε, ε, χρειάζονται λοιπόν στήριξη από πλευράς της Ευρώπης και αναγνώριση. Κατά τη γνώμη με αυτό το πρόγραμμα σημαίνει πως περνά και από την ενίσχυση των δικαιωμάτων και των αξιών της Ευρώπης. Και αυτό σημαίνει πρόληψη και αυτό σημαίνει ασφάλεια μεγαλύτερη. Αντίθετα, είμαι κάπως, ε, έχω κάποιες αμφιβολίες όσον αφορά τη δυνατότητα να μεταφερθούν πόροι στο πρόγραμμα ε, που αφορά τις περιπτώσεις παραβίασης του κράτους δικαίου. Ε, θα πρέπει να βρούμε εναλλακτικέ λύσεις που να μην ε, επιβαρύνουν εκείνους που στο εσωτερικό κάθε κράτος μέλος όπου μπορεί να υπάρξουν τέτοιες παραβιάσεις εργάζονται για την αποκατάσταση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας. Δηλαδή θα πρέπει νομίζω να συζητήσουμε και να προσπαθήσουμε να βρούμε συμβιβαστική σε αυτό το σημείο για να μην επιβαρυνθεί η κοινωνία των πολιτών. Ευχαριστήσω άλλη μια φορά την εισηγήτρια και είμαι πεπισμένη ότι θα εργαστούμε αρμονικά και με τους κοιόδης με ένα γρήγορο, ένα γρήγορο χρονοδιάγραμμα που θα μας επιτρέψει να ολοκληρώσουμε την εξέταση του προγράμματος εντός της θητείας αυτής. Ευχαριστώ. Um, e Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσουμε τον κύριο Γιούρεκ από το ECR. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το πρώτο το οποίο πρέπει να αποφασίσουμε είναι το εάν τα προγράμματα αυτά για τα οποία μιλάμε πραγματικά θα συνεισφέρουν σε κάποιες ε, δραστηριότητες ή σε κάποια ιδεολογία. Η κοινωνία των πολιτών σημαίνει κάποια δραστηριότητα την οποία μπορούμε να στηρίξουμε και με πόρους, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να στηρίξουμε συγκεκριμένες ιδεολογίες. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τις κυρίες Βαλέρο και Μίχαλ να ξεκαθαρίσουν την θέση τους. Η κυρία Μιχαλά ανέφερε, παραδείγματος χάρη, την ενδοοικογενειακή βία. Και θα ήθελα να γνωρίζω εάν με βάση αυτό το πρόγραμμα είναι δυνατόν να γίνει μια έρευνα για την βία στα ομοφιλόφιλα ζευγάρια. Εδώ μιλάω για, τον, ε, για προγράμματα του Διεθνούς συνασπισμού καταπολέμησης της βίας. Παραδείγματος χάρη με βάση αυτά τα προγράμματα ε, μπορούμε να μελετήσουμε την βία στα gay club. Στην ε, Πολωνία ακόμα και η γκαζέτα βιβότσα έχουν αναφέρει αυτό το πρόβλημα οπότε πρέπει να το λέμε. Οπότε το πρόγραμμα αυτό μπορεί να συνεισφέρει και σε κάποια έρευνα για την στήριξη οικογενειών πολυτεκνών. Γνωρίζουμε ότι αυτές οι οικογένειες αντιμετωπίζουν υλικά προβλήματα και πρέπει να τους ε, στηρίξουμε. Κάνω λοιπόν πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις. Δεν θέλω να ακούσω την απάντηση ότι όλα ε, στηρίζονται. Εγώ ρωτάω κάτι το πολύ συγκεκριμένο. Περιλαμβάνονται αυτά τα προγράμματα ή όχι. Σιλβί. Εσύ είσαι η αρμόδια εισηγήτρια. Θα ήθελες τον λόγο. Ε, με συγχωρείτε που ψίαζα ήμουν στην Επιτροπή Πολιτισμού για το θέμα αυτό. Η συζήτηση ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν από την Επιτροπή Πολιτισμού να συνεισφέρουμε με τον καλύτερο τρόπο σε αυτήν την έκθεση. Προφανώς θα έχουμε κάποιες ζώνες ε, επαφής όσον αφορά τον συντονισμό ε, μεταξύ μας. Για να δούμε ακριβώς ε, πώς θα οργανώσουν τη χρηματοδότηση της κοινωνίας, την επιπρόσθετη χρηματοδότηση της κοινωνίας των πολιτών. Γνωρίζω πως τελευταία είχαμε κάποιες τροποποιήσεις που αφορούσαν ακριβώς και το ύψος των χρημάτων ε, και την διαδικασία, αλλά δεν θα ήθελα να είμαι πιο λεπτομερής. Ε, ε, συνολικά τώρα θα τεθεί το θέμα ακριβώς ε, της αγωγής του πολίτη. Νομίζω ότι για το θέμα της ε, λέγης αυτής. Οπωσδήποτε θα γίνει μια συζήτηση για τα κονδύλια, το τι αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το τι πρέπει να φτιάξουμε. Και ακούγοντας τον κύριο Γιούρεκ με αυτές τις ερωτήσεις, ε, ε, νομίζω ότι στις εκθέσεις αυτές των δύο επιτροπών θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν κάποια τέτοια στοιχεία τι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει αποδείξει την χρησιμότητά του στον τομέα της αγωγής του πολίτη, της ε, χρησιμότητας των ΜΚΟ κτλ. Χρειάζεται ε, διευκρινήσεις και πρέπει να το στηρίξουμε με ε, επαρκή χρηματοδότηση στο μέλλον. υγιείς οργανώσεις της ε, κοινωνίας των πολιτών ε, αντιμετωπίζουν ε, θέματα πρόσβασης και εγώ είχα στο παρελθόν συζητήσει με τέτοιες οργανώσεις, γνωρίζω το θέμα. Η πρόσβαση αυτή τη στιγμή είναι συχνά πολύ δύσκολη. Και μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για δραστηριότητες θεμελιώδεις για τη δημοκρατία. Εκεί είναι οργανώσεις απαραίτητες για να έχουμε μια υγιή και δραστήρια κοινωνία των πολιτών. Και αυτές οι οργανώσεις βλέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύμμαχο. Δεν πρόκειται για μια προνομιακή μεταχείριση, αλλά για μια ίση μεταχείριση. Θέλετε και εσείς το... να απαντήσετε στα, στα σχόλια που έγιναν. Κύριε Μπόνι, ο Μάρεκ, ο συνάδελφός μας, μου έκανε μια ερώτηση και πρέπει να απαντήσω. Στο πνεύμα του διαλόγου, το πνεύμα είναι ανοιχτό. Αν μιλούμε για διακρίσεις, πρέπει κάθε φορά να αναλύουμε όλους τους τύπους διακρίσεων. Για κάθε ομάδα και χωρίς ταμπού. Οπότε, συμφωνώ μαζί σας. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε κάθε δραστηριότητα και σε κάθε ομάδα. Κάποιοι μπορούν να θεωρούν ότι πίσω από τα λόγια σας υπάρχει κάτι κρυφό, αλλά εγώ συμφωνώ με τη γενική διαπίστωση ότι θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε κάθε δραστηριότητα που είναι υπέρ της, των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπέρ της αξιοπρέπειας και κατά των διακρίσεων. Νομίζω ότι θα βρούμε τη λύση εκεί. Το πρόβλημα είναι για παράδειγμα όταν βλέπουμε τα ισχύοντα, τα τρέχοντα προγράμματα, προγράμματα βλέπουμε ότι έχουν πολλές σημαντικές δραστηριότητε που πρέπει να διατηρηθούν. Τι θέλουμε όμως τώρα. Θέλουμε να στηρίξουμε όχι μόνο τα ευρωπαϊκά διεθνή δίκτυα οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Όχι μόνο οργανώσεις κοινωνία των πολιτών που στηρίζονται από κυβερνήσεις με τη χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα καινούργια πυλώνα για τη στήριξη των οργανώσεων των πολιτών που έχουν ανάγκες και είναι σημαντικές για τη δημιουργία για την τροφοδότηση του διαλόγου στο πλαίσιο ενός τέτοιου διαλόγου καλό είναι να μην εξετάσουμε το θέμα με ιδεολογικές παροπίδες. Θα πρέπει να δούμε το θέμα αυτό σαν να είναι όλοι άνθρωποι, ίσοι άνθρωποι. Πρόεδρος Τζιν. Θέλεις να μιλήσεις? Ή για να απαντήσει σε κάποιον. Να, ζητώ συγγνώμη, αρχίζω να κουράζομαι. Η Τετάρτη είναι η καινούργια Πέμπτη. Κουράζομαι ήδη. Έχουμε ψηφοφορία στις 11.30. Παρακαλώ να είστε σύντομοι. Για να κάνουμε μία μικρή διακοπή πριν τις ψηφοφορίες 11.30. Είμαι εισηγήτρια στην ε, γνωμοδότηση της Επιτροπής ε, Απασχόλησης, οπότε θέλω να πω και εγώ δύο λόγια. Ε, σύμφωνα με τη συζήτηση που είχαμε και χτες στην Επιτροπή Απασχόλησης, δεν κοιτάξαμε το θέμα του προπολογισμού καθόλου. Το αφήσαμε για την αρμόδια, καθήλυνα αρμόδια επιτροπή. Ε, δεν έχω εντάξει ακόμα τις τροπολογίες στην νομοδότησή μου, αλλά να πω ποια είναι τα σχόλιά μας. Ε, πρώτον θέλουμε να μπει η λέξη ποιότητα στον τίτλο, ποιότητα και αρχές και αξία, συγγνώμη. Να προσθέσουμε δύο λόγια για το θέμα της καταπολέμησης των διακρίσεων, γιατί έχουμε και την οδηγία απασχόλησης για, που έχει σχέση με αυτό το θέμα. Επίσης το Equinet πρέπει να μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Ε, το Equinet προβλέπεται από την κοινοτική νομοθεσία με στόχο να προασπίσει τον ευρωπαϊκό νόμο, ποτέ έχει να παίξει σημαντικό ρόλο. Επίσης θέτουμε το θέμα του χώρου εργασίας. Είναι ένα καλό σημείο για να εργαστούν διάφορες ομάδες. Θέλουμε επίσης κάποιες τροπολογίες ε, και αντί να μιλάμε για πολίτες να μιλάμε για άτομα people στα αγγλικά Επίσης για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού ε, που είναι στερούνται συγκεκριμένων πόρων κλπ θα πρέπει αυτά τα προγράμματα να λειτουργήσουν σε συνέργεια με άλλα προγράμματα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπριγκέτε, έχεις να πεις μία φράση όμως μόνο. Έχω κάποιες πρόσθετες ερωτήσεις. 30 δευτερόλεπτα, αν μπορώ. Δύο-τρία ερωτήσει ακόμα. Υπάρχει το παράρτημα με τις ε, επιλέξιμες δράσεις. Ή μάλλον υπάρχει αυτή τη στιγμή τώρα στο καινούριο κείμενο όλες αυτές οι δράσεις μπαίνουν στο, στο ε, βγαίνουν από το παράρτημα, δεν υπάρχει πια παράρτημα και μπαίνουν στο σώμα. Δεν θα μπορούσα να ξαναμετακινηθώ σε παράρτημα. Δεύτερον, άρθρο για το διάλογο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κοινωνία των πολιτών. Αυτό είναι λίγο γενικόλογο ή οριζόντιο. Ίσως κάτι μου διαφεύγει για αυτό το καινούριο άρθρο. Τρίτον, γίνεται αναφορά στα εθνικά σημεία επαφή. Λένε ότι θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα. Λέγεται ότι θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα. Κάνα πρόβλημα. Ίσως όμως θα μπορούσαμε να δοθεί λίγο περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ που για την υπομονή σου, Μπρικίτ. Έχεις το λόγο. Κάνα πρόβλημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Δεν ε, θα ήθελα να πω κάτι για τις λεπτομέρειες ε, της πρότασης. Απλά θα ήθελα να πω πόσο επέσχυντο θεωρώ το ότι ε, συζητάμε καν τέτοια πρόταση εδώ στο Κοινοβούλιο. Γιατί υπάρχουν ανάλογα προγράμματα για χώρες εκτός της Ένωσης όπου θέλουμε να στηρίξουμε αξίες και δημοκρατία και τώρα μιλάμε για ένα τέτοιο πρόγραμμα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δυστυχώς αιτιολογημένα γιατί σε πολλά κράτη-μέλη και σε αυτά ε, τα οποία δεν είναι αυτή τη στιγμή ψηλά ψηλά στην ατζέντα μας, βλέπουμε ότι η δημοκρατία και το κράτος δικαίου, αλλά και οι αξίες όπως ορίζονται στην ε, συνθήκη, ε, κινδυνεύουν και εν μέρη ΜΚΟ οι οποίες εργάζονται για τη δημοκρατία και την μη διακριτική μεταχείριση δεν μπορούν να εργαστούν και είναι λυπηρό το ότι πρέπει να το συζητήσουμε όσον αφορά τις συγκεκριμένες ε, δραστηριότητες. Βεβαίω ε, εξαρτάται πάρα πολύ από κράτο μέλο σε κράτος μέλο, από περιφέρεια σε περιφέρεια, το τι θα γίνει, πού πρέπει να γίνει κάτι κτλ. Το θέμα του προπολογισμού είναι πραγματι δραματικό. Βλέπουμε και πάλι ότι στον τομέα αυτό λεφτά δεν υπάρχουν. Ε, συνάδελφος ή συνάδελφος ανέφερε ότι στον τομέα της δικαιοσύνης ε, υπάρχει μείωση, υπάρχει αύξηση σε άλλους ε, τομείς μεταξύ των οποίων στο Εράσμους, αλλά για να είμαι ειλικρινής και το Εράσμους δεν διευρύνεται, απλά μπαίνει εκεί το πρόγραμμα αυτό του Interrail. Οπότε δεν είναι περισσότερα τα λεφτά στο Εράσμους, ίσως να είναι και λιγότερα στη χειρότερη περίπτωση. Και ταυτόχρονα λέμε ότι τα κράτη-μέλη θα δώσουν περισσότερα λεφτά για στρατιωτικές δαπάνες. Εδώ πέρα κάτι πάει στραβά. Συμφωνώ επίσης με τον συνάδελφο Μπόνι ότι θα πρέπει να μην ε, μπούμε στην ιδεολογία, αν και βεβαίως εντάξει, ε, ο όρος αυτός είναι συζητήσιμος, το τι εννοεί ο καθένας. Επίσης αυτά τα οποία είπε ο κύριος Γιούρεκ επίσης είναι εξόχως ιδεολογικά όταν μιλάει για έρευνα σε γκέι κλαμπ, μιλάει για βία μεταξύ ομοφιλοφίλων ή κατά ομοφιλοφίλων. Ε, είναι κάτι το αξιοσημείωτο. Αλλά ε, η βία δυστυχώς ε, υπάρχει σε όλες τις κοινωνικές ομάδες και εξ όσων γνωρίζουμε και στην Καθολική Εκκλησία σε πολλά κράτη-μέλη. Και μια τελευταία παρατήρηση όταν μιλάμε για τη βία κατά των γυναικών. Δυστυχώς έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει εδώ, υπήρχε εδώ και αιώνες και δεν έχει ακόμα εξαλειφθεί και επειδή η μισή κοινωνία μας είναι γυναίκες είναι μια ιδιαίτερη πτύχη την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Σας ευχαριστώ Μπριγκίτε. Ηρέμησε λίγο η συζήτηση εκεί στο τέλος. Λοιπόν. Όλοι ε, θα μιλήσουν. Λοιπόν, Μπόντιλ. Να, ψηφι... να κάνουμε ένα διαλυματάκι γιατί σε λίγο θα έχουμε την ε, πιο μακροσκελή ψηφοφορία στην ιστορία της Επιτροπής μας. Οπότε, παρακαλώ, σύντομα τα συμπεράσματά σας. Σας ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη. Έγιναν κάποιες ερωτήσεις ε, για το θέμα αυτό της αγωγής του πολίτη. Προτείναμε μια αλλαγή στον ε, τίτλο γιατί είναι ένα θέμα το οποίο ετέθη από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ε, και όταν θέλουν Ε, να παραμείνει κάτι. Εμείς θεωρήσαμε λοιπόν ότι θα πρέπει να τονίσουμε τη λέξη πολίτης εδώ πέρα. Κάτι ευρύτερο από την έννοια της ηθαγένειας, υπηκότητας κτλ. Οπότε ε, αυτό προτείναμε. Δεν μπήκε ο τίτλος ισότητα, αλλά μπορεί να γίνει μια τροπολογία. Συμφωνώ με την Σεσίλ ότι πρέπει να περιληφθεί αυτό το οποίο είπε για συγκεκριμένα μέτρα τώρα. Ε, θα πρέπει να το δούμε στο πρόγραμμα εργασία ε, ή το τι θα μπει συγκεκριμένα στο νομοθετικό κείμενο. Και νομίζω θα πρέπει να περιληφθούν και οι οργανώσει κοινωνία των πολιτών στι διαβουλεύσεις ε, του προγράμματο εργασία για να εγκριθεί δηλαδή το πρόγραμμα εργασία. Τώρα, αρκετοί ανέφεραν τα σημεία επαφή, αν είναι κάτω θετικό ή αρνητικό. Υπάρχουν κάποια σημεία επαφή που λειτουργούν πολύ καλά για κάποια προγράμματα και με αυτή τη βάση το κάνουμε αυτό. Όλοι θα πρέπει να έχουν ένα εθνικό σημείο επαφής, αλλά πρέπει να είναι ανεξάρτητοι ε, και να ισχύει αυτό για όλα τα προγράμματα. Αλλά ευχαρίστως να δεχτώ οποιαδήποτε πρόταση για βελτίωση. Και νομίζω τελικά θα καταλήξουμε σε μια λογική λύση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νομίζω είναι Ε, είναι ενδεικτικό το ότι ασχολούμαστε τόσο πολύ με μια πρόταση του προϋπολογισμού και πολλές ε, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών παρακολουθούν. Οπότε ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ και τους κοιόδης συγητές. Λοιπόν, συναδελφοί ψηφοφορία θα ξεκινήσει 11.30. Να έχετε τις κάρτες σας. Κάνουμε ένα διάλειμμα λίγων λεπτών. Θα ξεκινήσουμε 11.30 ακριβώς. So, dear colleagues, please um, be ready. Um, it's all electronic as usual. I always say this particularly for the substitute members. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσουμε γρήγορα ε, με τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες για τέσσερις εκθέσεις. Ορισμένες, ε, ε, ε αυτή που σίγουρα που έχει να κάνει με το Facebook είναι κάπως περίπλοκη, γι' αυτό... Ε, θα πρέπει να προσέξουμε όλοι πολύ. Πρώτη έκθεση, ε, Πάβελ, εδώ νομίζω ψηφίζουμε σχεδόν για όλα. Εκεί λίγο να προσέξετε. Ε, ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη ψηφοφορία που είναι η έγκριση του σχεδίου έκθεσης που θεσπίζει την Ευρωπαϊκή Αρχή Ε, εργασίας ε, εισηγητής ο κύριος Εμίλιαν Πάβελ. Λοιπόν, ξεκινάμε με ε, τις ψηφοφορίες. Τροπολογία 20 άρχεται. Τέλος. Απορρίπτεται 75. Άρχεται. Απορρίπτεται 76. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται 77. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. 78. Άρχεται. Τέλος. Απορρίπτεται. 79. Άρχεται. Τέλος. Καλά. 80 άρχεται. Τέλος. Απορρίπτεται. 81 άρχεται. Closed. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. 82. Άρχεται. Τέλος. Απορρίπτεται. 83. Άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. 84. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. 85. Τέλος. Απορρίπτεται. 86. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. 87. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8 ψηφίζουμε. Τέλος. Εδώ οι σοσιαλιστές είχαν ένα παραπανίσιο βουλευτή που ψήφισε. Οπότε παρακαλώ ένας από εσά να βγάλει την κάρτα του. Εντάξει τώρα. Ωραία λοιπόν εγκρίνεται. Τροπολογία 89. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 9. Άρχεται. Τέλος. Ε, εγκρίνεται. Τροπολογία 90. Τέλος, εγκρίνεται 10 Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. 91. Τέλος. Απορρίπτεται. 92. Τέλος. Έγκρινεται. Τροπολογία 11. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. 93. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. 94. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. 95. Τέλος. Απορρίπτεται. 13. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. 96. Τέλος. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 4. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. Εκατόν δύο. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. 103. Ψηφίζουμε. Απορρίπτεται. 104. Απορρίπτεται. 105. Άρχεται. Τέλος. Απόρριπτεται. 106. Τέλος. Εγκρίνεται. 107. Τέλος. Εγκρίνεται. 108. Τέλος. Απορρίπτεται 109. Τέλος. Απορρίπτεται. Συμβεβαστική τροπολογία 5. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. 112. Άρχεται. Τέλος. Απορρίπτεται 113. Άρχεται. Τέλος. Απορρίπτεται 114. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται 115. Ψηφίζουμε. Τέλος εγκρίνεται 116 ψηφίζουμε τέλος εγκρίνεται 118 ψηφίζουμε τέλος εγκρίνεται 119 ψηφίζουμε Τέλος. Εγκρίνεται. 120. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. 16. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. 121 ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. 122 ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. 17 ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. 18. Ψηφίζουμε. Τέλος. Έγκρινεται. 19. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. 125. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. Εκτιμώντας 21, ε, όχι έχει αποσυρθεί, πάμε σε θεολογικές σκέψεις, τροπολογία 22 άρχεται, τέλος, απορρίπτεται, 23 άρχεται, τέλος, εγκρίνεται. 24 Δεν μπορούμε δυστυχώς να κάνουμε μπλοκ, λυπάμαι, πρέπει να πάμε μία-μία. Τις απολογίες. εγκρίνεται λοιπόν, 25 ψηφίζουμε. Δεν έχουμε συνηθίσει τέτοιου είδους ψηφοφορίες, εν πάση περιπτώσει Τέλος ψηφοφορίας τώρα. Απορρίπτεται. 26. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. 27. Τέλος. Εγκρίνεται 28. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται 29. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται 30. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται 31. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. 32. Τέλος. Εγκρίνεται. 33. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. 34 ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. 35. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. 36. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. 37. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1. Τέλος. Εγκρίνεται. Πάμε λοιπόν στην τροπολογία 2. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. 42. Τέλος. Απορρίπτεται. 43. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. 44 ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 2 άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 48. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. 49 ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. 50. Τέλος. Απορρίπτεται. 51. Τέλος. Απορρίπτεται. 52 ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. 53 ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. 54 ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. 55 ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. 57 ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. 58 Τέλος. Απορρίπτεται. 59. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. 60. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. 61. Α, όχι, 62. Ε, ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. 63. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. 64. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. 65. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. 66 ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 71. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. 72. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. 73. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. 74. Ψηφίζουμε. Τέλος. Αν κρίνεται. Και τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Ψηφίζατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται με 39 ψήφους υπέρ, 7 κατά και 4 αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Okay. Ωραία. Τώρα περνάμε στο δεύτερο θέμα. Ελάχιστα πρότυπα για τις μειονότητε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγητής ο Γιώζεφ Νάζ. Θα ήθελε το λόγο. Όχι, πάμε κατευθείαν στη ψηφοφορία. Ετοιμή. Τροπολογία υπαριθμών 3. Σημαντική τροπολογία υπαριθμών 3. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 94. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 95. Μόνο το δεύτερο τμήμα. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Πολλοί μιλάνε εκεί στο ΕΛΚΑ, αλλά τέλο πάντων. Συμβαστική τροπολογία 4. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 177. Λήξη. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία υπερθυμών 6. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7. Έναξη. Στη σελίδα 24. Ψήφισατε όλοι. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8. Σελίδα 20 κύριε Μπέκερ. Τροπολογία 289. Λήξη. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 9. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 10. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1 στα εκτιμώντας. Έναρξη. Είναι στη σελίδα 40 του δικού μου καταλόγου. Λήξη. Συμβαστική τροπολογία 2. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 76. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 82. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Πολύ μικρή διαφορά. Προσέξτε λοιπόν. Τελειώσαμε. Ψηφίζουμε το κείμενο στο σύνολό του. Έναξη ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Λήξη. Εγκρίνεται 44 ψήφοι υπέρ, 4 κατά, 4 αποχές. Συγχαρητήρια στον κύριο Νάτζ. Ωραία. Αυτή ήταν... Ε, αυτός ήταν κατάλογος ψηφοφοριών. Λοιπόν, εδώ πέρα θα καθαρίσουμε λίγο γιατί είναι κάπως πιο πολύπλοκο. Η χρήση δεδομένων των χρηστών του Facebook από την Cambridge Analytica και ο αντίκτυπος στην προστασία των ε, δεδομένων. Να ευχαριστήσω όλες τις πολιτικές ομάδες ε, για την στήριξή τους ε, και για τις ακροάσεις που ήταν δύσκολο να στηθούν. Ψηφοφορία στην Ολομέλεια, στην δεύτερη Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Λοιπόν, θα πάω πιο σιγά εδώ. Κύριε Βος, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα εξ ονόματος του, ΟΛΚ να κάνω, του ΕΛΚ να κάνω μια σύντομη δήλωση. Στο τέλος αυτού του ψηφίσματος θα υπερψηφίσουμε, αλλά οπωσδήποτε δεν θα δεχτούμε αυτήν την τροπολογία για το Privacy Shield και σας παρακαλώ να δεχτείτε να μην την συμπεριλάβετε, αν και στο τέλος έχουμε βάλει ένα σύν όπως σας είπα. Το σημειώσαμε κύριε Βος, δεν σας αρέσει πράγματι, κατανοητό. Είστε ευγενικό και θα το ψηφίσετε στο τέλος. Όμως, είστε πολύ ευγενικοί. Δεδομένου του ότι αυτή είναι η θέση τώρα, ας μην το συζητήσουμε. Γι' αυτό ακριβώς ε, θα πάω λίγο πιο σιγά γιατί υπάρχουν κάποια αιτήματα για ονομαστική ψηφοφορία από το ΕΛΚ, οπότε ας ε, το δούμε λίγο πιο προσεκτικά. Ξεκινάμε με την 29. Άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρασε. Απορρίπτεται. 30. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 32. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τώρα περνάμε... Εντάξει, σας παρακαλώ λίγο συγκεντρωθείτε. 33. Άρχεται τη ψηφοφορία. Ε, εντάξει, δεν θέλω να σου πω αλλά είναι δύσκολη ψηφοφορία. 33. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 34. Άρχεται τη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 35. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρας απορρίπτεται 36 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 37 άρχεται ψηφοφορία πέρας δεκτή 38 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 41 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 44 όχι. 42 συναδελφοί. Πέρας. Δεκτή. 44 αρχιτιψοφορία. Πέρας. Δεκτή. 45 αρχιτιψοφορία. Πέρας Πέρας. Απορρίπτεται. 46 έξι, αρχιτεί ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 48 οχτώ, αρχιτεί ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 49 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Δεκτή. 51 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 52 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 53 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 54 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 55 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. απορρίπτεται. 56 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Τόμας, είσαι εντάξει. Ωραία. Απορρίπτεται. 57 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην 61 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 62 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 63 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 64. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 65 έρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 66 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Δεκτή. 60 71. Έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 74. Όχι, 72. Έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 74 αρχιτή ψηφοφορία. Πέρασε. Δεκτή. 75 μέρος πρώτο αρχιτή ψηφοφορία. Πέρασε. Δεκτή μέρος δεύτερο αρχή ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 76 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 77 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 78 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 79. Άρχιδη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 80. Άρχιδη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 81. Άρχιδη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 82 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 83 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 84 αρχιτή ψηφοφορία. Πέρασε. Δεκτή. 86 αρχιτή ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 87 έχουμε ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησε το ΕΛΚ, αρχιτή ψηφοφορία ονομαστική. Πέρας. Δεκτή. Μπράβο, Άξελ. 88. Άρχεται η ψηφοφορία. Γι' αυτό ελέγχουμε τα πάντα σε αυτή την επιτροπή. Πέρας. Απορρίπτεται. 89 άρχεται η ψηφοφορία. Δεκτή. 90 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Πέρασε. Δεκτή. 92 αρχή η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 93 αρχή η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 94 αρχή η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 95 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 96 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 97 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας δεκτή 98 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται ε, κάνουμε και την 99 άρχεται η ψηφοφορία πέρας δεκτή εκτιμώντας 1 άρχεται η ψηφοφορία Πέρασε. Κάνουμε όλα μαζί. Ωραία. 2 έως 6, 2 έως 7. 2 έως 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Δεκτά όλα. Τώρα περνάμε στα εκτιμώντα. 8 και 9 μαζί. Άρχεται η ψηφοφορία. Α, όχι. Δεν γίνεται. Α, συγγνώμη. Μπορούμε. Μπορούμε. Πέρασε. Απορρίπτονται και τα δύο. Δέκα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 11 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Δεκτή. Ναι, δεν γίνεται. Λοιπόν, 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 14. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε. Δεκτή. Δεκαπέντε. αρχιτή ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Δεκαέξι. άρχιτη ψηφοφορία. Πέρασε. Δεκτή. 17 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 18. Άρχεται η ψηφοφορία και πέρας. Απορρίπτεται. 19 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Η 20 άρχεται. Πέρας. Αδεκτή. Συμβιβαστική 1 αρχιτή ψηφοφορία. Πέρας. Αδεκτή. 21 αρχιτή ψηφοφορία. Ναι. Σωστά. 21 μέχρι 28. Όχι. Όχι, 21 μέχρι 26 και μετά περνάμε στον Άξελ Φως. Ωραία, 21 μέχρι 26. 21, άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρασε. Καλή προσπάθεια, Μπίργκιτ. Απορρίπτονται. 22 άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. 23 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 25 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 26 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 27 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 28 άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρας. Και απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Δεκτή με 41 ψήφους υπέρ, 10 κατά και μία αποχή. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Άλλη μία έχει μείνει. So let's, go, let's just get to it fast, colleagues, and then we'll, it'll be over. Να την τελειώσουμε και αυτή γρήγορα γρήγορα. Ανθρωπιστικές θεωρήσεις, θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους. Φερνάντο Λόπε Αγγιλάρ, ο εισηγητή. Θέλει το λόγο πριν περάσουμε στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν ψηφίζουμε μια έκθεση την οποία την έχουμε δουλέψει τόσο πολύ καιρό και έχουμε βρει συμβιβασμούς, είναι χρήσιμο να ευχαριστούμε τους και ηγητές ε, για την ικανότητά τους να καταλήξουν σε αποδεκτούς συμβασμούς. Αυτή η έκθεση προσπαθεί να είναι συνεπής με τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτές που έχει υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ευαίσθητα θέματα. Ξεκινώντας από την έκθεση με τσόλα, την ολιστική αποκαλούμενη προσέγγιση του μεταναστευτικού προβλήματος και χαίρομαι που το Κοινοβούλιο κατέληξε σε μια τόσο κοινή θέση. Προσπαθούμε να στείλουμε ένα μήνυμα ιδιαίτερα στα πιο ευάλωτα άτομα, αλλά και προς την Κομισιόν και προς το μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους προσπάθησαν. Okay, thank you very much, Juan. Πρόεδρος, κύριος Μπέκερ, ο ηγητής για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. αρκετά κάποια μέλη της ομάδας μου ε, δεν θα ακολουθήσουν τη σύστασή μου να ψηφίσουν υπέρ. Θέλω να διευκρινίσω ότι η απόφαση να υπερψηφίσουμε προκύπτει από έναν συμβασμό της ΣΑΛΤΕ που υιοθετήθηκε από τον εισηγητή. Οι ανθρωπιστικές θεωρήσεις δεν θα είναι υποχρεωτικές για τα κράτη-μέλη πλέον και από την άλλη μεριά αντιλαμβανόμαστε ότι η σχετική έκθεση για τον κώδικα περί θεωρήσεων των αναδιατυπωμένων ε, μετά από ε, προσπάθειες της γραμματείας και του εισηγητή άλλαξε και το καινούριο χρονοδιάγραμμα μας επιτρέπει να προχωρήσουμε επιγόντως και να ολοκληρώσουμε το φάκελο κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας συμπεριλαμβανομένων και των τριμερών διαλόγων που θα ξεκινήσουν φέτος. Θέλω να εμπιστευτώ αυτό το κοινό χρονοδιάγραμμα. Θέλω να πιστέψω ότι θα τηρηθεί και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, και όλοι οι και όλα τα μέλη, έτσι ώστε αυτή η έκθεση να αποτελέσει μια επιτυχία. Ο κ. Μωρέσης, είναι ευαίσθητο το θέμα. Υπάρχουν εκκρεμή θέματα, προφανώς ελπίζω ότι ε, μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 1. Άρχεται. Λίγη. Ε, εγκρίνεται. Τροπολογία 74. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 157. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Ονομαστική έναρξη. Λήξη. 39 ψήφοι υπέρ, 10 κατά. Καμία αποχή. Συγχαρητήρια στον εισηγητή και στους κοιόδης. Ευχαριστώ πολύ συνάλφοι για την υπομονή σας. να καταφέραμε. Τέλος της πληροφορίας.